Colleagues, please take seat. We Καθίστε συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Our economic dialogue. Να ξεκινήσουμε διάλογο, να καλωσορίσουμε την Υπουργό από την Πορτογαλία, την κυρία Μαριζάλ Μπουκέρκη. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Υπουργό Επικρατεία και Οικονομικών τη Πορτογαλίας για να συζητήσουμε την κατάσταση στην Πορτογαλία, μια χώρα που όπω γνωρίζετε τον Ιούλιο του 2014 βγήκε και επισήμως από το πρόγραμμα οικονομική προσαρμογή και μετά από μια σταδιακή επιστροφή στις κεφαλαιαγορές, από τον Ιούλιο του 2014 η Πορτογαλία πλέον έχει ε, ενταχθεί πλήρως στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στο πλαίσιο της ε, δημοσιονομικής μακροοικονομικής εποπτείας. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Μοσκοβισή μας παρουσίασε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού των κρατών μελών και η Πορτογαλία συγκαταλέγεται μεταξύ των ε, χωρών που η ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κινδυνεύει να μην συμμορφούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία την ίδια ημέρα να συζητήσουμε την κατάσταση στην Πορτογαλία, την οποία θα μας παρουσιάσει η Υπουργό Αλμπουκέρκε και να σας δώσω απευθείας το λόγο για την παρουσίαση της κατάστασης. Παρακαλώ. Thank you, President. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σε αυτή την πρώτη ακρόαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ, Οικονομικών και Νομισματικών, λίγους μήνες μετά την ε, προσαρμο, το πρόγραμμα προσαρμογής της Πορτογαλίας έχει τεράστια σημασία να επισημάνουμε ποιες είναι οι κυριότερες πρόοδοι που έγιναν καθώς επίσης και τις προκλήσεις που υπάρχουν ακόμη. Το πρόγραμμα προσαρμογής ε, συνελήφθη για να επιληθούν τα διαθωτικά προβλήματα της ε, οικονομίας μας και ξεκινήσαμε το 2011. Από τα μέσα της δεκαετίας ε, του 90 και λόγω της προετοιμασίας για το ευρώ και λόγω της μη τήρησης κάποιων αρχών υπήρξαν μεγάλες ε, μη ισόρροπες σχέσεις ε, στην Πορτογαλία και την οικονομία της. υπήρξε γενική χρέωση, υπερχρέωση του κράτους των επιχειρήσεων της ίδιας της χώρας εναντί του υπόλοιπου του κόσμου και παράλληλα η ανάγκη να οικοδομηθεί μια οικονομία πιο ανοιχτή και πιο ανταγωνιστική ε, εξετάστηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ε, μια μεγάλη περίοδος ε, αποτελμάτωσης που οδήγησε σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, ιδιαίτερα ευάλωτη μέσα στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Τον Απρίλιο 2011 με την κατάρρευση του διεθνούς πλαισίου το, ε, ε, η ε, ανάγκη για την προσαρμογή της οικονομίας μας ήταν κάτι αδύρυτο ανάγκη είχαμε κυριότερες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Δημοσιονομική εξυγίανση για την ε, αηφορία των δημοσίων οικονομικών. Συνεργασία όσον αφορά την σταθερότητα. Διαρθρωτικές αλλαγές για την αηφορία στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σήμερα μετά την ε, ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής η αποτίμηση είναι θετική είχαμε την δυνατότητα να μειώσουμε το έλλειμμα από το 11,5 σε 4,9 το 2010 και καταφέραμε να έχουμε από το 1997 την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την διαρθρωτική προσαρμογή κατά 6 μονάδες. Και έτσι προχωρήσαμε το 2014 όπως δείχνουν τα στοιχεία μας. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση η δημοσιονομική και η φορολογική έδωσαν τη δυνατότητα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεγαλύτερης διαφάνειας. Συνεισφέραμε για μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων λογαριασμών. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σημείο ως Μετά από δεκαετίες ελλημάτων καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2013. Στο δημοσιονομικό πλαίσιο καταφέραμε να συνδεθούμε με τις χρηματοδοτήσεις των αγορών και ποτέ ε, ε, δεν, σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Είναι μια μακροπρόθεσμη προοπτική και διατηρούμε τις επαφές ε, με την οικονομία της αγοράς και η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Ξεκίνησε μια γενική διαδικασία καθώς επίσης και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που αύξησαν τη δυνατότητα των τραπεζών να μπορέσουν να αντισταθμίσουν απώλειες και έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρχουν πιστώσεις ε, για την οικονομία. Διαρθρωτικά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα που ήταν ευρύτερων ε, διαστάσεων για την οικονομία μας που είναι πιο ανοιχτή και πιο δυναμική δημιουργώντας ε, ε, πλεονεκτήματα που θα έχουν αηφόρο παράμετρο. Η ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής έκανε αναγκαία την αποτίμηση. Να δούμε ποιοι τομείς χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Σε αυτή τη σύντομη περίοδο που είναι μεταβατική περίοδος θα πρέπει να δούμε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης οδήγησαν σε ε, πάρα πολλά μέτρα τα οποία ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των τριών ετών. Το πρόγραμμα αυτό ε, έχει νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο διαθωτικό τομέα έχουμε ένα νέο ε, χάρτη που έχουμε ε, δημιουργήσει στην ε, οικονομία μας. Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της ΤΑΠ των εναέριων μεταφορών της Πορτογαλίας ξεκίνησε απλά και μόνο για να δώσω τα πιο συμβολικά παραδείγματα. Η σφαιρική προσπάθεια προσαρμογής άνοιξε τον δρόμο, τον δρόμο για την δημιουργική οικονομική δραστηριότητα σε τριμηνιαία επισκόπηση είχαμε ανάπτυξη που από τότε συνεχίζεται. Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία εξετάσαμε δείχνουν μια ανάπτυξη η οποία συνεχίζεται κατά το δεύτερο εξάμεινο και έχουμε 1% ε, ποσοστιαίας μονάδας ε, αύξηση της ε, οικονομίας μας. Με αηφόρο τρόπο συνεχίζεται ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 4,4% και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαμε κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους την, την αναλογική αυτή αύξηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυξητική πορεία. Το πρόγραμμα προσαρμογής έδωσε την δυνατότητα να επανορθωθούν ε, οι μη ισόρροπες σχέσεις που υπήρχαν στην αγορά. Όμως υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε και με σθένος ε, αντιμετωπίζονται κατά τα τελευταία τρία έτη. Ήταν αποφασιστικές οι πρόοδοι που σημειώθηκαν, όμως ε, τα προβλήματα που ε, παρουσιάστηκαν το 2011 δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Πρέπει ακόμα να αναμείνουμε ε, στο εγγύς μέλλον την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων επανόρθωσης οι δείκτες σε σχέση με τα όρια μακροοικονομικά δείχνουν την ε, καθαρή θέση ρευστότητας ε, και το επίπεδο σε σχέση με το ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας ήταν τα πρώτα σημεία τα οποία αναλύθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες ε, για την ε, ε, αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους και του ελλείμματος. Υπάρχει ακόμα ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια προσαρμογής ώστε να δημιουργηθούν βάσεις αιφόρες, Το ποσοστό της ανεργίας συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες και μεγάλο κόστος προσαρμογών. Και πρέπει σε σχέση με το 2010 να πούμε ότι η ανάγκη ήταν κατεπίγουσα το 2011 και ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης στην οικονομία που οδήγησε στην αύξηση μέχρι την αρχή του 2013 του ποσοστού ανεργίας στην Πορτογαλία. Υπάρχει ακόμα μια άλλη πρόκληση και που πρέπει να αναγνωριστεί ακόμα ε, ε, δεν είναι μόνο η ανάγκη των ε, μη ισορροπών σχέσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά πρέπει μέσα στο οικονομικό πλαίσιο να αντιμετωπιστούν όλες οι ανάγκες. Τα προβλήματα της οικονομίας μας έκαναν να δράσουμε με κατεπήγοντα τρόπο. Σήμερα η προσαρμογή έχει και πάλι κατεπήγοντα χαρακτήρα και πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε βάσεις αηφορίας για την οικονομία ιδιαίτερα όσον αφορά το πλαίσιο το οποίο, στο οποίο θέλουμε να κινηθούμε. Η σημασία αυτού, αυτής της ε, ισορροπίας είναι σαφής για το 2015. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ε, μετά το πρόγραμμα προσαρμογής αλλά έχει και σημασία συμβολική. Γι' αυτό τον λόγο ε, ξεκινήσαμε έγκαιρα μέσα στο πλαίσιο του στρατηγικού, των στρατηγικών εγγράφων για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει καθοριστεί η δημοσιονομική προοπτική ε, μεσοπρόθεσμα, αλλά έχουν εντοπιστεί και τα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ε, επίτευξη του ορίου του, ε, της, υπερχρέωσης, της χρέωσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος και την αντιμετώπιση ε, του υπερβολικού ελλείμματος. Και έτσι είδαμε σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό εγχείρημα τα δημοσιονομικά έτη 2014-2015. Αυξήθηκαν οι δυσκολίες με το νέο σύστημα λογαριασμών που άρχισε να ισχύει. Σαν αποτέλεσμα τα μέσα της εξυγίανσης ε, που είχαν αρχικά υιοθετηθεί δεν επαρκούσαν για να υλοποιηθεί το αναγκαίο ποσοστό για το έλλειμμα το 2015 σε σχέση με τους διεθνείς μας εταίρους. Συνολικά ταυτοποίησε μέτρα εξυγίανσης η κυβέρνηση ε, όσον αφορά το ε, 0,7% του ΑΕΠ. Έδινε τη δυνατότητα αυτό να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, αλλά δεν ήταν επαρκές αυτό για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η πρόκληση συνολικά που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία. Ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων δαπανών σε σχέση με τις δράσεις για την ανάπτυξη θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς μια πολιτική συνένεση από τον πολιτικό κόσμο. Λήφθησαν λοιπόν τα αναγκαία μέτρα για ε, την προσαρμογή των δαπανών και θεωρήθηκε ότι η υπερβολική φορολόγηση θα ήταν αντιπαραγωγική δράση. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θέλει να διασφαλίσει το 2015 την έξοδο της Πορτογαλίας από το ε, μνημόνιο και την ε, ε, συνεχή της πορεία. Όμως υπήρξαν και θετικές εξελίξεις όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα καθώς επίσης και τα δημοσιονομικά. Συνεχίζουμε με μόνιμο χαρακτήρα να επιτηρούμε την κατάσταση ώστε έγκαιρα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας στις ανάγκες, αν χρειαστεί αυτό. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, οι μεταρρυθμίσεις ε, που ε, υιοθετήθηκαν στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δημιούργησαν τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη δυνατότητα εφορία. Ωστόσο, η τροχιά αυτή θα πρέπει να απαιτήσει συνέχεια των προσπαθειών και οι προκλήσεις είναι εξίσου σημαντικές και η ευθύνη είναι αυξημένη όσον αφορά την δράση μας. Έχει συνειδητοποιήσει η κυβερνήση της Πορτογαλίας ότι δεν είναι χωρίς κινδύνους αυτή η πορεία, ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι είναι η σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ξεκινήσουμε με τον γύρο των αγοριτών. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο κύριος Γιώργος Χρήστος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αφού πρώτα συγχαρώ την Υπουργό, γιατί πιστεύω ότι η Πορτογαλία τα, τα πήγε πολύ καλά, τα πηγαίνει καλά, γιατί στο κάτω-κάτω μπήκε στο πρόγραμμα μετά την Ελλάδα, τη χώρα μου, και βγήκε με αρκετά καλές επιδόσεις πριν από εμά. ήθελα να της κάνω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο έχει σχέση με την έξοδο στις αγορές. Σε ποιο βαθμό έχει βγει το πορτογαλικό δημόσιο στις αγορές. Δηλαδή, καλύπτει ε, παίρνει κάποια χρήματα για να συμπληρώσει τα χρήματα του προγράμματος που φτάνουν στο τέλος τους ή έχει την εμπιστοσύνη των αγορών και μπορεί και δανείζεται με αρκετά χαμηλά επιτόκια οπότε κάνει αναδιάρθρωση του χρέους και γλιτώνει, δηλαδή περιορίζει το κόστος της διαχείρισης του χρέους. Αυτό ήθελα το πρώτο. Ε, και το δεύτερο είναι ένα πρακτικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και ήθελα τη γνώμη της και τη συμβουλή της. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που κρίνουν αντισυνταγματικές μειώσεις συντάξεων και μισθών, για παράδειγμα των δικαστικών λειτουργών, των αστυνομικών, ίσως ακολουθήσουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου και οι γιατροί του Δημοσίου. Επομένως υποχρεώνεται η κυβέρνηση και δίνει πίσω τα λεφτά που είχε πάρει στα πλαίσια του προγράμματος και παίρνει αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι δυσάρεστα και αντιπαραγωγικά, όπως η αύξηση του ΦΠΑ στο ξενοδοχειακό τομέα που είναι ανταγωνιστικός τομέας για την Ελλάδα. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό, γιατί ξέρω ότι είχατε κι εσείς δικαστικές αποφάσεις που σας υποχρέωναν να δώσετε πίσω τα χρήματα που είχατε πάρει από το πρόγραμμα λιτότητας. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Το θέμα της εξόδου στην αγορά μετά το τέλος του προγράμματος ήταν μια εναλλακτική λύση που συνεπαγόταν κινδύνους. Όμως κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών η Πορτογαλία κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και κατάφεραμε να περάσουμε στις αγορές αυτό το μήνυμα ότι δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και προσπάθεια της κυβέρνησης και της χώρας για να αντιμετωπιστούν τα διαθέτικα προβλήματα και να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα είναι πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας και που θα είχαμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε το χρέος μας και να προχωρήσουμε σταδιακά σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες αλλά επίσης και όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η αυξημένη αξιοπιστία από πλευρά μας είναι εκείνη που μας οδήγησε στο να καταφέρουμε στα πρώτα βήματα να αρχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στις αγορές με την αναγκαία εμπιστοσύνη και δεν χρειάστηκε κανένας μηχανισμός υποστήριξης πέρα από το ότι είχαμε δημιουργήσει ένα απόθεμα ρευστότητας για την αντιμετώπιση σχετικά μακρότερων περιόδων ε, λόγω ευμετάβλητου χαρακτήρα των αγορών για να μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, συνταγματικές αποφάσεις. Στην Πορτογαλία πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είχαμε κάποιες αποφάσεις, κάποιες συμφωνίες του συνταγματικού δικαστηρίου, κάποιες αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου που παρα παρακόλλησαν την υλοποίηση μέτρων που είχαν αποφασιστεί από την κυβέρνηση και δεν συνεχίστηκαν. Και αυτό οδήγησε στο να αλλάξει η κατανομή, ο επιμερισμός των προσπαθειών μας όσον αφορά τις δαπάνες. Στο αρχικό πρόγραμμα είχαμε μια δυνατότητα των δύο τρίτων όσον αφορά τις δαπάνες να υπήρχε μια, ε, ένας περιορισμός και αντιστάθμιση από πλευράς εσόδων και στο συνολικό πρόγραμμα έπρεπε να γίνει μια ε, ε, ανακατανομή μισό-μισό, 50-50, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την εξυγίανση όσον αφορά την ε, κατάσταση αυτή. Όμως το πλαίσιο το συνταγματικό είναι αυτό το οποίο είναι και οι αποφάσεις και η νομολογία του συνταγματικού δικαστηρίου είναι αυτές που είναι και έχουμε ως κυβέρνηση το καθήκον να σεβόμαστε τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου και να υιοθετούμε τα μέτρα εκείνα τα οποία επιτρέπεται για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους μας. Δεν είναι τα καλύτερα μέτρα αυτά γιατί αν θα μπορούσαν να ήταν τα καλύτερα θα τα είχαμε λάβει ήδη την πρώτη φορά χωρίς την τροποποίησή τους. Ωστόσο ήταν ε, αντιληπτό ότι υπήρχαν Έγιναν αυτές οι, ε, αυτοί οι περιορισμοί, σεβαστήκαμε τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου και υιοθετήσαμε άλλα μέτρα, τα οποία μας επέτρεψαν ακόμα και έτσι να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Ευχαριστώ. Κυρία Λίζα Φερέιρα από τους Σοσιαλδημοκράτες, καλώς ήρθατε σε αυτή την κοινοβουλευτική μας επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο. Κυρία Υπουργέ, ήδη γνωρίζουμε εμείς ότι εμείς θέτουμε σε αυτή τη διαδικασία διαφορετικές απόψεις έχουμε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η κυβέρνηση που επομίζεται τις ε, διοικητικές ε, ε, ευθύνες και από πλευράς Υπουργού Οικονομικών ήταν πάντα ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις θέσεις και απόψεις της Τρόικας και ακόμα και πέρα από αυτές. Αναγνωρίζουμε τα στοιχεία τα οποία συναποτελούν την αρχική αυτή προσπάθεια και τη, για τη μείωση του χρέους, ε, διαθωτικές αλλαγές ε, και μεταμόρφωση της, οικο, της οικονομίας μας ε, και δημοσιονομικά μέτρα. Σήμερα έχουμε ένα κείμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου εξετάζοντας την Πορτογαλία αναγνωρίζεται ότι το ιδιωτικό χρέος είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Παραβιάζονται λοιπόν τα όρια που έχουν τεθεί μέσα στο scoreboard των πίνακα επιδόσεων. Και έτσι λοιπόν είναι 128 το χρέος μας. Πάλι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Εξεράγει η, το ποσοστό ανεργίας. Έχουμε μια κατάσταση για τις επενδύσεις που είναι πολύ αρνητική. Χάσαμε ποσοστά αγορών όσον αφορά τις εξαγωγές μας. Και έχουμε και μια κατάσταση όπου έχουμε ε, μιλιάδες ε, ανέργους ε, πάμπολους ε, μετανάστες νέους, όλα αυτά αφέμαξη της οικονομίας μας. Στην ανάλυση που κάνουμε, αν, κάνοντας μια επισκόπηση προς το παρελθόν, προσπαθώντας να αντιληφθούμε τι δεν πήγε, καλά στην διαδικασία προσαρμογών, η δική σας συνεισφορά θα ήταν πάρα πολύ σημαντική σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή ακόμα και το θέμα του ελλείμματος θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως μη αηφόρο, μη ε, βιώσιμο. 3,3% του ΑΕΠ πρέπει να ήταν. Έχουμε ήδη παραβιάσει το ε, όριο. Και κατηγορείται η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ότι βρίσκεται σε μια παρεκκλίνουσα ε, πορεία. Υπάρχει ή δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα σε σχέση με τη σωστή πορεία. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Βλέποντας προς τα πίσω και την προοπτική που εξετάζουμε, κάποια πράγματα θα ήθελα να είχαν συσταθεί και να είχαν ακολουθηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η συνταγή της Τρόικας όμως ε, έπρεπε να γίνει σεβαστή. Υπήρχαν όμως δυνατότητες ε, ίσως να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε γι' αυτό κάτι. Και όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα διαρθρωτικής εξυγίανσης και παγίωσης, τι θα προτείνατε εσείς Υπουργέ για να, υλοποιηθεί, να υλοποιηθούν ή όχι οι συστάσεις της Επιτροπής για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτή και για το ότι με καλωσορίσατε. Το ότι πήγε πιο πέρα από την Τρόικα και η κυβέρνηση είναι κάτι το πολύ, πολύ συζητημένο στη χώρα μας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να πούμε είναι ότι έχουμε απόλυτη συνδυτοποίηση της ανάγκης επανόρθωσης των μεγάλων ανισοτήτων και μεγάλων ε, μη ανα, ε, ισόρροπων σχέσεων που υπήρχαν στην Πορτογαλία. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο και που χρησιμοποιήθηκε το ότι ο όρος, η έκφραση πήγαμε και πιο πέρα από την, ε, τις συστάσεις Τρόικα. 12 Ωστόσο, η αντιμετώπιση του χρέου, η δυνατότητα δημιουργία θέσεων απασχόληση και εξυγίανση των δημοσιονομικών πράγματι έχει σοβαρό πρόβλημα η Πορτογαλία, διότι συσσωρεύονται, συσσωρεύθηκαν τα προβλήματα. Η Ιρλανδία έχει πρόβλημα ιδιωτικού χρέου, για παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει χρέο, δημόσιο χρέο. Η Πορτογαλία έχει και δημόσιο χρέο και ιδιωτικό χρέο, ε, που είναι, ε, δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση. Και γι' αυτό έπρεπε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιλύσουμε το πρόβλημα ε, ε, το, του στόκ πέρα από το, το θέμα των ε, ε Και θα έπρεπε να γίνει μια μακρόχρονη προσπάθεια για να μπορέσει να ανατραπεί μια κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα σε μια περίοδο πάνω από μια δεκαετία. Δεν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει εν μια νυχτή λοιπόν. Το δημόσιο χρέος είναι 128% όμως το ιδιωτικό χρέος είναι 118% που παρόλα αυτά δημιουργεί μια διαφορά και σε σχέση με τις ε, εξαγωγές μας ε, δεν έχουμε χάσει τόσα πολλά. Έχουμε ε, επανέλθει στις αγορές, σε πολλές από τις αγορές που είναι σημαντικές για μας και καταφέραμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αγορές. Έχουμε πολυμορφοποιήσει και κάνει πιο πολυσχηδή τις δράσεις μας σε σχέση με τον ευάλωτο χαρακτήρα τους κατά το παρελθόν, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το έλλειμμα για του χρόνου, έχουμε μια διαφορά ε, μεταξύ μας των προβλέψεων. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι λογικές οι δικές της προβλέψεις. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σε σχέση με την ε, πρώτη συλλογή μετά την, ε, το μνημόνιο δείχνει ότι σε σχέση με το 2014 έχουμε βελτιώσει τα πράγματα. Με πρόσθετα μέτρα θεωρούμε δεν θα έπρεπε να υιοθετηθούν πρόσθετα μέτρα τα οποία θα επιβάρυναν την οικονομία μας και θα ήταν αντιπαραγωγικά. Και γι' αυτό λέμε δεν πρέπει να τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα και θα χρησιμοποιήσουμε επαρκώς ε, τις δυνατότητες ε, ανάπτυξης που έχουμε και θα είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας αν καταστεί αναγκαίο. Έχουμε απόλυτη ασθεναρή δέσμευση που έχουμε αναλάβει να αντιμετωπίσουμε το χρέος και το έλλειμμα. Ευχαριστώ. Μα ήταν μία η ερώτησή μου. Η διαδικασία προσαρμογής ακολουθήθηκε νέου ή τι συνέβη με αυτήν. Ευχαριστώ. Κυρία Ευρωβουλευτά, η ερώτηση που θέσατε, εγώ ε, ακολούθησα τη σειρά των παρατηρήσεών σας ε, στην απάντησή μου. Εν πάση περιπτώσει, Απλά και μόνο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπήρξε η ανάγκη να γίνουν προσαρμογές κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Έγιναν αυτές οι προσαρμογές. Ήταν μια διαδικασία μάθησης ε, αυτή για τα όργανά μας ε, όσον αφορά προσδοκίες του πληθυσμού μας που ήταν τελείως διαφορετικές. Ε, και έχουμε και μια ολόκληρη διαδικασία αναδιάρθρωσης που ήταν μάθηση για μας. Κανονικά πάντα θα ήταν δυνατό να πει κανείς ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα. Όμως πήγαμε καλά και αντιμετωπίσαμε τα πιο κατεπήγοντα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις σαφείς ε, απαντήσεις. Ε, έχασα λίγο την αρχή της ομιλίας σας, γιατί έπρεπε να είμαι σε άλλη επιτροπή. Θα ήταν πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Πορτογαλία, αλλά και για σας ε, να πούμε το εξής. Τώρα, λόγω του προγράμματος Golden Visa Investment, ήταν στις ειδήσει η Πορτογαλία. Αυτό ε, είναι ένα μεταξύ παρομοίων επενδυτικών προγραμμάτων ε, ή δεν είναι έτσι. Στη Λετωνία έχουμε και εμείς ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Αυτό αφορά περισσότερο την ε, ε πώληση ε, ηθαγένειας στο χώρο του Σέγγεν. Μια τέτοια επένδυση σε μια αγορά καταστρέφει... Α, είναι ε, πώληση ε, κατοικιών ε, στο έδαφος του Σέγγεν και αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι τιμές και στη Λετωνία λιγότερο από ό,τι στην Πορτογαλία. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τα δημοσιονομικά. Το Golden Visa επενδυτικό πρόγραμμα πώς το κρίνετε στη χώρα σας και σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν παρόμοια προγράμματα. Ακόμα και αν τα διαχειρίζονται καλά συμβάλλουν σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και δεν υποσκάπτουν την ασφάλεια. Επίσης πιστεύετε ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να παραμείνουν ε, επιχειρησιακά μακροπρόθεσμα ή μόνο βραχυπρόθεσμα μέσα στην κρίση και μετά να σταματούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το, το, πρόγραμμα Golden Visa σε ποιο βαθμό στρεβλώνει τα επενδυτικά πρόγραμμα σε χώρες όπως Πορτογαλία, Κύπρο, Μάλτα και άλλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτά. Πράγματι το πρόγραμμα αυτό σε σχέση με τα όσα αναφέρονται με βάση οι ειδήσει ε, που ίσως δεν είναι απόλυτα ορθές, όμως ε, στο σωστό του πλαίσιο όσον αφορά το ίδιο το πρόγραμμα υπάρχουν πραγματικά παρόμοια προγράμματα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που πάνε πιο πέρα από αυτό το οποίο ε, δίνεται κιόλας και η ηθαγένεια μέσω αυτών και όχι μόνο η άδεια παραμονής. Εμείς από ό,τι είδαμε με αυτό το πρόγραμμα αδειών παραμονής έδωσε τη δυνατότητα να αναζωογονηθούν τομείς των ακινήτων, της αγοράς ακινήτων που ε, βρέθηκαν σε στασιμότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και λόγω των διαστάσεων της αγοράς μας ή λόγω της επιτυχίας του προγράμματος δεν είναι αυτό γνωστό σε όλους. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδαμε και συναντήσαμε είναι μια ανάκαμψη της αγοράς των ακινήτων που είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και δεν είδαμε κάποια στρέβλωση που να συνδέεται με αυτή την ανάκαμψη στα ακίνητα. Παράλληλα είχαμε και επενδύσεις σε άλλους τομείς επενδύσεις για παράδειγμα σε ε, ταμεία, σε αποθεματικά και είδαμε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου για να επαληθεύσουμε την προέλευση αυτών των κεφαλαίων είναι πάρα πολύ αυστηροί και επιτυγχάνεται η συνεργασία χρηματοοικονομικών τομέων της αστυνομίας των διοκτικών αρχών από διάφορες χώρες. Έχουμε ένα πολύ σύνθετο ε, σύστημα ε, αλληλοδιάδοχων επαληθεύσεων και ελέγχων για την προέλευση αυτών των κεφαλαίων ώστε να μην επιτρέψουμε να είναι ε, φεά τα κεφάλαια τα οποία θα εισέρχονται. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για την Πορτογαλία είναι ότι αυτό το πρόγραμμα συνεισέφερε για την αναζωγόνηση της αγοράς και την εισφορά, την εισαγωγή κεφαλαίων και την δυνατότητα ε, νέων την, νέες δυνατότητες που άνοιξε στον τραπεζικό μας τομέα. Και σε σχέση με τις ε, στρεβλώσεις που ε, αναφέρατε δεν υπάρχει κάποιος ορίζοντας προβλέψιμος για να τερματιστεί αυτό το πρόγραμμα. Πάντα βρίσκεται σε διαρκή αξιολόγηση και τι Εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών μέσω ελέγχων και σε σχέση με αυτή την επιτήρηση που είναι διαρκής θα μπορούμε πάντα να προσαρμόσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποιους αντικειμενικούς λόγους για να υπάρξει απόφαση να, τερματιστεί αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Next speaker, Η επόμενη Μαρίζα Ματίας από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Υπουργέ. Η κυβέρνηση λέει ότι το πρόγραμμα προσαρμογής ήταν επιτυχία λέει. Μια τοποθέτηση αυτού του είδους δεν μπορεί να γίνεται με βάση τις αξιολογήσεις της Τρόικας. Μια σοβαρή αξιολόγηση απαιτεί να δούμε τους στόχους του προγράμματος ε, αυτού προσαρμογών με τα αποτελέσματα και να δούμε στο 2014 τι υπάρχει σε σχέση με το μνημόνιο και τι θα συμβεί σε σχέση με το ΑΕΠ. Ε, είχαμε μείωση κατά 5 και παραπάνω τα 100. Η απασχόληση μειώθηκε και αυτή. Το ποσοστό ανεργίας ε, αντί 12% είναι 14%. Έλλειμμα θα έχουμε αντί 3% 4%. Και βλέπουμε ότι η αποσταθεροποίηση τώρα σε σχέση με το χρέος είναι 128% του ΑΕΠ. Αποτέλεσμα, σε όλες τις παραμέτρους υπήρξαν παραβιάσεις και επιδεινώσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν είχε σαν, στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες ε, στη χώρα, πώς είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση που είναι επιδείνωση να θεωρείται επιτυχία. Δεύτερη ερώτηση σήμερα είχαμε μία τοποθέτηση πολύ σοβαρή ε, του Επιτρόπου Μοσκοβίση ότι η Πορτογαλία δεν τηρεί τα συμπεφωνημένα και ότι θα είναι πολύ στενή η παρακολούθηση, η εποπτεία της Πορτογαλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότι ακούστηκαν και κάποια αισιόδοξα πράγματα. Καταφέρατε να δημιουργήσετε προβλήματα λέγοντας ότι θα αντιμετωπίζατε τα προβλήματα. Ακολουθήσατε τις συστάσεις της Τρόικας. Είδαμε ότι τα προβλήματα της χώρας επιδεινώθηκαν, δεν βελτιώθηκαν αυτό που είδαμε σε σχέση με, την, τα όσα αναφέρθηκαν είναι ότι έχει υποστεί την τιμωρία, τις ποινές που, έπρεπε να, ε, που, επιβλήθηκαν σε αυτήν η Πορτογαλία. Αρχίζει μια πολεμική αντιπαράθεση, μια ε, διαφορά και σύγκρουση μεταξύ ε, των θέσεων της κυβέρνησης και των επιχειρημάτων της. Είδαμε ότι έχασε όλους τους στόχους η κυβέρνηση ακολουθώντας τις συστάσεις της Τρόικας. Τώρα όμως υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβλημα και για αυτό το ζήτημα θα ήθελα να μου πείτε εσείς πρώτα απ' όλα παρακολούθησα τον κανονισμό όσον αφορά τα τραπεζικά ότι όλοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι προτού ε, θεωρηθεί ότι πρέπει οι φορολογούμενοι να επομιστούν τις απώλειες. Και όταν είδαμε ότι οι απώλειες μετακυλίστηκαν σε εκείνους που δεν έφταιγαν να τις ε, επομιστούν. Αντί λοιπόν ε, να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι ε, αγνοώντας και τις αρχές του κοινοτικού δικαίου και με την Τράπεζα της Πορτογαλίας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολιτικές είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Και η δεύτερη πτυχή, αν όπως αναγνωρίστηκε από τους διάφορους υπεύθυνου, θα υπάρξουν απώλειες για τους φορολογούμενους, είτε άμεσα ή μέσω της, της Γενικής Τράπεζας ε, του Γενικού Ταμείου Αποθεματικών, τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα έβαιναν Σε Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτά. Έμεινε όμως πολύ λίγος χρόνος για την απάντησή μου. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε σχέση με αυτά τα οποία ήταν προβλέψεις και αυτά που συνέβησαν, αν επαληθεύσετε τις προοπτικές και προβλέψεις για όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης και συγκρίνετε με αυτό το οποίο πραγματικά συνέβη, θα δείτε ότι τα σφάλματα για τις προβλέψεις δεν είναι αποκλειστικό, αποκλειστικά κάτι το οποίο επιβαρύνουν την Πορτογαλία. Έγιναν και αλλού τέτοιες ε, ε, διαφορές, υπήρξαν και αλλού τέτοιες διαφορές όσον αφορά τις προβλέψεις. Ιδιαίτερα όταν είχαμε τέτοια θέματα προσαρμογών. Αυτό είναι που είναι σημαντικό για την Πορτογαλία είναι να πούμε, να δούμε αν υπήρχαν άλλες αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις. Η απάντησή μας είναι όχι, δεν υπήρχαν. Ακολουθήσαμε αυτή την πορεία, τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Δεν είναι ακριβώς αυτοί οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί. Όμως βρισκόμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, πιο αηφόρα και έχουμε στοιχεία θετικά για όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Δεν έχει κάτι αυτό το οποίο είναι δογματικό, είναι πράγματι πεποίθηση. Πεποίθηση ότι ήταν τεράστια η συσσόρευση ε, διαρθωτικών προβλημάτων και τεράστιο πρόβλημα η αντιμετώπιση τους. Και έπρεπε λοιπόν πραγματικά να πούμε ότι βρεθήκαμε σε μια τραγική κατάσταση. Κοινωνική κοινωνικά και οικονομικά με τεράστιες επιπτώσεις. Όσο αφορά το ερώτημα που θέσατε για τις διαφορές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της κυβέρνησής μας, εμείς έχουμε μια κατάσταση μη υλοποίησης υποχρεώσεων των συμπεφωνημένων. Επειδή όμως θεωρούμε ότι οι δικές μας ε, προβλέψεις δεν, έπρεπε, δεν ε, πρέπει να τροποποιηθούν ε, άρδιν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σταδιακή προσαρμογή, γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πέρα από το ότι σε σχέση με την Πορτογαλία οι αποφάσεις για τους μηχανισμούς αυτούς που ελήφθησαν έδιναν προοπτική αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ένα ελάχιστο burden sharing, επιμερισμός βαρών για τους ε, μεριδιούχους και ομολογιούχους. Ε, και πρέπει να πούμε ότι αυτό θα, είναι, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο προστασίας των φορολογουμένων. Υπάρχει λοιπόν δεδομένη ευθύνη για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Αν υπάρξει μια ολόκληρη σειρά γεγονότων που ε, δημιουργεί μια ξεχωριστή κατάσταση για την Casa Gerard de αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα Άντε. Παραμένει η τέταρτη ε, ομάδα. Τόρβατ παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ε, πάντοτε δίνουμε πρώτα το λόγο στις κυρίες. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας κυρία μου. Συναντηθήκαμε σύντομα κατά τη διαδικασία με την Τρόικα όταν σας επισκεφθήκαμε στο Υπουργείο σας. Σήμερα ε, εξετάσαμε κάποια θέματα μακροοικονομικών ανισορροπιών και τα στοιχεία για την Πορτογαλία, όπως είπατε, έχετε ποσοστό ανεργίας ε, μεγάλο, ε, κίνδυνος φτώχειας υψηλός επίσης. Ας υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, πάρει το πρόγραμμα αυτό των 300 δις και ότι εσείς ε, θα πάρετε το μερίδιο που σας αναλογεί από εκεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματά σας, αυτές οι επενδύσεις που πρέπει να διοχετευθούν για να είναι όσο γίνεται αποτελεσματικότερες. Γιατί αν δεν βαθμονομήσουμε τις επενδύσεις αν θέλετε μπορεί να υπάρξει διασπάθηση χρήματος πράγμα καταστροφικό, καταστροφικό για μας και πιθανόν και για σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Αλήθεια είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε κατά το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ήδη ήταν πολύ υψηλός ο κίνδυνος αυτός και πριν από το πρόγραμμα και το ίδιο ισχύει για την ανεργία. Πράγμα που δείχνει ότι αυτό που έκανε η κρίση είναι να αναδείξει προβλήματα που είχε εδώ και καιρό η Πορτογαλία. Δηλαδή δεν τα φτιάξε η κρίση, απλώς αποκαλύφθηκαν μέσα από την κρίση. Και αυτό σκοπό έχει να δείξει ότι στην πραγματικότητα είχαμε μπροστά μας τεράστιο έργο γιατί έπρεπε να διορθώσουμε μα παλιές ανισορροπίες σε διαφόρων διαστάσεων μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και την Ευρώπη που ήταν σε βαθιά κρίση και ποτέ δεν είναι εύκολο να επιλύεται ε, η εσωτερική κρίση. Αυτό ήταν το περιβάλλον που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Κατόπιν τούτου πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να διορθώνουμε τις ε, ανισορροπίες για να μειώνουμε το ποσοστό φτώχειας που είναι, τον κίνδυνο φτώχειας που είναι πολύ ψηλός. Πάρα πολύ ψηλός. Ποια άλλα όμως ρεαλιστικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν για να μειωθεί αυτό το ποσοστό βραχυπρόθεσμα. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, συνέχιση των προσπαθειών για την διόρθωση των διαρθρωτικών ανισορροπιών για να μην, και να μην έχουμε την ψευδέστηση της στιγμιαίας μεγέθυνσης ανάπτυξης αλλά κάτι διατηρήσιμο που θα μπορέσει να ε, ε, κρατήσει τα νούμερα αυτά χαμηλά. Όχι να λύσουμε τεχνητά το πρόβλημα και μετά από δύο χρόνια να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή τις προσπάθειες και πιο επώδυνες. Πρέπει να δούμε ποιο ήταν το σημείο εκκινήσεως της Πορτογαλίας και ποια είναι τα προβλήματα που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Παρόλο που οι δείκτες βελτιώνονται ήδη, ακόμα εξακολουθούμε να έχουμε πολλά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Τώρα για το πρόγραμμα Juncker. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό για μας, όχι μόνο για τις επενδύσεις που θα γίνουν στην Πορτογαλία, αλλά και σε σχέση με ευρωπαϊκές επενδύσεις που θα έχουν σχετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά μας. Συνεχίζουμε να ε, τονίζουμε την σημασία της δημιουργίας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Για μια χώρα περιφερική όπως είναι η Πορτογαλία είναι πολύ σημαντικό, είναι θέμα κλειδί για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, οι τιμές ενέργειας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού τομέα παραγωγής μας. Και αν τμήματα αυτού του επενδυτικού πακέτου πάνε προς αυτό το στόχο, ακόμα και χωρίς τις άμεσες επενδύσεις, θα είναι όφελος. Θα ωφελήσει όλη την ε, ε, ζώνη του ευρώ. Θα είναι ε, ωφέλιμο και για την Πορτογαλία προφανώς. Αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι ιδιωτικέ επενδύσεις. Έχουμε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα έλλειψη κεφαλαίων στο, στις επιχειρήσεις μας. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Υπάρχει υπερμόχλευση στις ε, επιχειρήσεις, υπάρχει θέμα ε, μετοχικού κεφαλαίου, αλλά χρειάζεται εισρωή κεφαλαίου, ιδίων κεφαλαίων, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή ε, από το χρέος στις, στα ίδια κεφάλαια. Χρειαζόμαστε γι' αυτό ιδιωτικές επενδύσεις. Όποια κεφαλαιακά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουμε την πρόοδο ε, στο σχεδιασμό μέσων που θα αντιμετωπιστούν το χρέος ε, και τις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά, όλα αυτά χρειάζονται για τη χώρα. Και είμαστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε όφηση και στην Ευρώπη και η Πορτογαλία θα ωφεληθεί από αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Μόρλιν Σκοτ Κέιτον από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξέταζα και εγώ τους μακροοικονομικούς δείκτες και πρόσεξα ότι τα στοιχεία του ισολογισμού έχουν βελτιωθεί. Οι μικρές βελτιώσεις όμως έγιναν με κοινωνικό κόστος, δηλαδή μείωση δημοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών επιδομάτων κλπ. Επίσης, ο λόγος χρέους ΑΕΠ δεν βελτιώνεται. Ο λόγος αυξήθηκε στα χρόνια του προγράμματος προσαρμογής και αυτό μου δείχνει ότι απέτυχε το διορθωτικό πρόγραμμα προσαρμογής. Είναι σαφές ότι το μεγάλο δημόσιο χρέος ε, δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα και πώς επιμερίζεται μεταξύ πολιτών και δανειστών. Πιστωτών. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτον, μπορείτε να μας πείτε το συνολικό αντίκτυπο του δημοσίου χρέους της Πορτογαλίας ε, και ε, για τη διάσωση ε, του δημοσιονομικού τομέα, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επίσης οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν τόσο πολύ για ένα δημόσιο χρέος το οποίο είχε να κάνει με την κοινωνικοποίηση ιδιωτικών απολειών και ζημιών. Επίσης η διαδικασία ελέγχου ποια θα είναι ούτως ώστε να κατανοήσουν και οι πολίτες πώς έγινε αυτό το χρέος, πώς ισορρεύθηκε και ε, αν η αναδιάρθρωση είναι ή δεν είναι ε, σωστή εναλλακτική. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι όντως ε, υπάρχει πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος, αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι προσαρμογές ε, έπρεπε να γίνουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ε, υπήρχε ε, πρόβλημα χρηματοδότησης και η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει έλλειμμα. Χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση ούτε ιδιωτικών ούτε δημοσίων κοφαλιών θα υπήρχε αμέσως κατάλληλος ολογισμός στον προπολογισμό, αλλά το κοινωνικό κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο για τους πολίτες. Επομένως η λύση δεν ήταν μεν εύκολη ε, και φυσικά ήταν επώδυνη για πολλούς πολίτες μας, αλλά ήταν σίγουρα καλύτερη λύση από την εναλλακτική λύση που είχαμε αντιμετωπίσει και που θα είχαμε αντιμετωπίσει σε περίπτωση που δεν υπήρχε μνημόνιο και δεν υπήρχε και δυνατότητα ε, να έχουμε χρόνο να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις και να ανακτήσουμε αξιοπιστία και πρόσβαση στις αγορές. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών έχει διατηρηθεί. Έχουμε ακόμα ένα ε, πολύ καλό εθνικό σύστημα υγείας, έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης, η ε, χώρα μας εξακολουθεί να είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο και στην Ευρώπη φυσικά και είναι μια καλά λειτουργούσα ε, χώρα. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν καταλήλως και κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εξορθολογήσουμε το κόστος, διότι πραγματικά αυτό θεωρούμε ότι χρειάζονται οι πολίτες, να μπορούμε να παρέχουμε την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και να διαγράψουμε οποιοδήποτε κόστος δεν χρειάζεται ε, για να μπορέσουμε να παρέχουμε κατάλληλης ποιότητας υπηρεσίας. Οι συνέπειες της διάσωσης του οικονομικού τομέα τώρα. Θα ήθελα να πω ότι από τις ε, τράπεζες που χρειάστηκαν ε, κρατική παρέμβαση μία έχει ήδη πλήρως αποπληρώσει ε, το χρέος της και το κόστος των επιτεχείων που καθορίστηκαν από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, ήταν πάρα πολύ καλή πηγή εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η δεύτερη τράπεζα έχει επιστρέψει το μεγαλύτερο τμήμα της στήριξης και ε, εξακολουθεί να είναι ε, στο σωστό δρόμο για την πλήρη επιστροφή. Υπάρχει μία δημόσια τράπεζα, αλλά επειδή ακριβώς είναι δημόσια εμείς είμαστε οι μέτοχοι και ε, υπάρχει μια σύγχυση εδώ μεταξύ του ρόλου των μετόχων και του ρόλου του κράτους εδώ και οι μεταβατικές αυτές επενδύσεις θα επιστραφούν και έχουν εξυπηρετήσει και το σκοπό τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι συνολικά το, ότι το κόστος για το κράτος και τους φορολογουμένους για τις παρεμβάσεις στον οικονομικό τομέα στην Πορτογαλία είχε θετικό αντίκτυπο. Ε, ξέρουμε όλοι ότι ε, χρειάστηκε να διασώσουμε μια τράπεζα το Δεκέμβριο του 2014, μετά το πέρας λοιπόν του προγράμματος. Ε, το κόστος αυτής της παρέμβασης απαιτεί ε, δάνειο, ε, δανειοδότηση από το ε, κρατικό κορβανά, αλλά θα είναι δάνειο και επειδή έχουμε ακολουθήσει τους κανόνες δεν θα υπάρχει κανένα κόστος για τους φορολογουμένους. Όσον αφορά τον έλεγχο των πολιτών για το χρέος, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί πιστεύουμε στη δημοκρατία. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν και να κατανοούν ε, και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ε, και να είναι ένα απόσπαστο τμήμα των αποφάσεων που λαμβάνονται και σε προεκλογικές περιόδους αλλά όχι μόνον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το χρέος είναι μνήμη. Είναι μνήμη των περασμένων χρεών, των περασμένων προβλημάτων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η μνήμη, ώστε τα σφάλματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Εξακολουθώ να λέω λοιπόν ως Υπουργό Οικονομικών ότι το χρέος είναι εκεί από το οποίο θα πρέπει να αντλήσουμε τα περισσότερα διδάγματα, διότι θα πρέπει να αντικατανοήσουμε τι πήγε στραβά, ποιε ήταν οι σωστέ αποφάσει, ποιε ήταν οι λανθασμένε αποφάσει και να διαβεβαιωθούμε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη απόφαση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Επομένω, μαθαίνουμε από τι προηγούμενε αποφάσει Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από το EFTD, επομένως τώρα να δώσουμε το λόγο στην Βάρμπαρα Κάπελ. Από τη ε, έχουμε πλέον ε, το λόγο για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να γίνει ένας ε, διάλογος για την οικονομική πολιτική. Εσείς ε, συνεχίζετε την ε, πολιτική του προκατόχου σας, του κυρίου Κασπάρ, για την εξηγίαση του προϋπολογισμού, μείωση χρεών, ε, διασφάλιση σταθερότητας δημοσιονομικής, δημιουργία ανάπτυξης με βάση τις προδιαγραφές της Τρόικα. Και αν δούμε τους μακροοικονομικούς σας δείκτες, πρέπει να πούμε ότι σε τρεις τομείς, το 2014, σε τρεις τομείς έγινε μια σημαντική αλλαγή ε, και στις επενδύσεις και στην εγχώρια ζήτηση. Το 2014 έχετε αύξηση του ΑΕΠ από 0,9 ε, ε, που είναι υψηλότερο από τις ευρωζώνης και του χρόνου προβλέπεται 1,3. 5,3 υψηλότερο από τις στις ε, η χώρια ζήτηση ε, αυξήθηκε περισσότερο από την Ευρωζώνη και στις επενδύσεις του 1,1 και 0,6 Ευρωζώνη. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ υπήρξε μια πολύ μεγάλη ε, αλλαγή και τον Ιούνιο φέτος μπόρεσε να ξαναγυρίσει στις κεφαλαίες αγορές με λογικά επιτόκια και να ε, γίνει επιτυχώς ο δανεισμός. Ε, κάνατε διαρθρωτικές αλλαγές που δημιούργησαν συμπάθεια για τη χώρα σας και βεβαίως το, ε, δημιούργησε και προβλήματα και δυσαρέσκεια, υπόθηκε αυτό σήμερα. Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την πορτογαλική οικονομία, φαίνεται ότι ακολουθεί ανωδική πορεία. Πώς κρίνεται σήμερα τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα λιτότητας. Πιστεύετε ότι ήταν σημαντικά για να γίνει ξανά η Πορτογαλία ανταγωνιστική. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτά. Πρωτού απαντήσω στην ερώτησή σας, απλά και μόνο να πω ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2014 η πρόβλεψη της κυβέρνησής μας ήταν 1%. Και για το τρίμηνο έχουμε 1,1% και μέρος ε, της ε, διαφοράς ε, με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για το πώς θα ολοκληρωθεί το 2014 και γι' αυτό οι διαφορές που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμεί ευελπιστούμε ότι η δική μας πρόβλεψη είναι πιο κοντά σε εκείνο το οποίο θα επαληθευτεί και βλέπουμε, προβλέπουμε για το επόμενο έτος 1,5% προς το ανάπτυξης μπόρεσε να ανακάμψει σε αυτή την πορεία ανάκαμψη η, η Πορτογαλία ιδιαίτερα σε σχέση με μια διαδικασία που είχε σταματήσει και μάλιστα σε πορεία σύγκλησης με τη ζώνη ευρώ και το ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αν υπάρχει κάποια διαφορά δεν είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εργαστούμε ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Καταφέρνουμε να μειώσουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της κατάσταση της Πορτογαλίας και της κατάστασης των άλλων χωρών χωρών ζώνη ζώνης ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως ε, προαναφέρθηκε. Εκείνο το οποίο αναφέρεται στις διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων που υλοποιείται και τελεία και παύλα ολοκληρώθηκε. Πρέπει να ε, συνεχιστεί και να συνεχίσουμε να σταθμίζουμε και να αποτιμούμε το τι γίνεται στην εξέλιξη αυτών των δράσεων. Έχουν κέρια σημασία. Πρέπει να συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Έχουμε κάνει πολλά. Πρέπει όμως να βελτιωθούν ε, οι διαδικασίες αφορά την ελαστικότητα, την ελαστικοποίηση μορφών εργασίας στην αγορά εργασίας. Και πρέπει η, ε, το επίπεδο ικανοτήτων να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς από πλευράς των εργαζομένων, Πορτογάλων εργαζομένων. Και είναι ένα χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό, όχι μόνο πορτογαλικό. Δηλαδή να πάψει να υπάρχει ο κατακαιρματισμός και να μπορέσει να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα με γνώσεις, με δεξιότητες, με ικανότητες. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα ε, ε, στοιχείων που πρέπει να οδηγήσουν ώστε να μπορέσουν να ε, εξηγιανθούν τα οικονομικά μας, τα δημοσιονομικά μας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία έχουν επιπτώσει στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας ε, με μια αηφόρο δράση, με αηφόρες δράσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα το θέμα των συντάξεων, το συνταξιοδοτικό, που πρέπει με μια διευρυμένη συνένεση να να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά η δημογραφική κατάσταση της χώρας μας ε, καθιστά αναγκαία το να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε τις διαθωτικές αλλαγές που χρειάζονται. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομολητής, Ιβάν Μάλεβιτς, ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ εδώ να καλωσορίσω την Υπουργό Οικονομικών της ε, Πορτογαλίας. Με χαρά διαπίστωσα ότι η κυβέρνηση της Πορτογαλίας και η Υπουργό Οικονομικών είναι στο σωστό δρόμο και υλοποιούν τους στόχους της οικονομικής πολιτικής για το 2015 ήδη η δημοσιονομική εξυγίανση και η ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτό είναι αυτό το οποίο ε, λέει σε όλα τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη στον προπολογισμό σας. Έχετε καταφέρει να αυξήσετε την ανάπτυξη και να μειώσετε τις άλλες δαπάνες. Οι συνάδελφοι σας έθεσαν ε, πολλές ερωτήσεις για το σχέδιο επενδύσεών σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ξέρω εγώ είναι ε, ποια είναι τα βασικά προβλήματα για την αύξηση των επενδύσεων στην Πορτογαλία. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκές ε, κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα. Εκ παραλίλου όμως υπάρχει πρόβλημα και με την καινοτομία, ίσως την παιδεία, ή ε, την πολύ περίπλοκη διοίκηση. Ποιες πηγές χρηματοδότησης έχετε στις οποίες δεν αναφερθήκατε ίσως και με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να επιλύσετε όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά ε, σχετίζονται στα, με τα 400 μέτρα τα οποία δηλώσατε ότι θέλετε να ελοπίσετε. Όσον αφορά τον τομέα της χρηματοδότησης ε, για τους επιχειρηματίες, αναφερθήκατε ε, στα equity instruments και στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου έπρεπε να καθοριστούν ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πτωχεύσουν διότι ήταν υπερχρεωμένες. Υπάρχει ε, κατάλογος πλέον αυτών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευρωβουλευτά. Σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξη του προϋπολογισμού μας 2015. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια ανάκαμψη των εισοδημάτων, οικογενειακών εισοδημάτων. Έχουμε την ε, απάλληψη μια σημαντική εισφοράς όσον αφορά τις συντάξεις ε, πάνω από 1000 ευρώ διατηρείται μόνο μια συνεισφορά αλληλεγγύης ε, σε σχέση με τις πιο αυξημένες συντάξεις έχουμε μια ανάκαμψη όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την αντιστάθμιση για την, ε, τις ε, ε, περικοπές που είχαν γίνει και έχουμε και μια μεταρρύθμιση του, της φορολόγησης εισοδημάτων που ανοίγει δυνατότητες ε, για τις ε, ε, οικογένειες που με παιδιά ιδιαίτερα σε σχέση με μια χώρα με χαμηλή δημογραφική ανάπτυξη που πρέπει να μπορέσει να συνεισφέρει για την επίλυση αυτού του προβλήματος και που με, χρόνο με χρόνο που περνάει καθίσταται όλο και πιο επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του. Έχουμε και μια δυνατότητα πράσινης φορολόγησης να ανακατευθυνθεί η παραγωγή για πιο αηφόρους περιβαλλοντικά. Να προσπαθήσουμε κάποιες τρευλώσεις που υπάρχουν εις βάρος του περιβάλλοντος στην αγορά να τις αντιμετωπίσουμε. Ο προϋπολογισμός όμως δεν ήταν ακόμα δυνατόν να περιορίσει τη φορολογία, τους φόρους. Και θα μπορέσουμε το ποσοστό φορολόγησης από 23% να μειωθεί σε 21% σε σχέση με μια μεταρρύθμιση που είχαμε αρχικά σχεδιάσει το 2011 για να υπάρξει μια καλύτερη, ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επενδύσεις. Έχουμε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμα οι επιχειρήσεις μας σε αυτόν τον τομέα. Σε κάποιους τομείς έχουμε θέματα που συσχετίζονται με το εργατικό δυναμικό και την ανάγκη να ε, μπορέσουμε μπορέσουν να γίνουν οι προσαρμογές. Έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες καινοτομίας και κατάρτισης για το εργατικό μας δυναμικό, εξαιρετικά, ε, εξαιρετικές ε, ευκαιρίες που προσφέρονται και σε σχέση με άλλες ε, χώρες έχουμε βελτιώσει ε, ε, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με αποτέλεσμα, αποτελέσματα αξιοπρόσεκτα και πραγματικά και στον επιστημονικό τομέα και επιχειρησιακό τομέα έχουμε σημαντικές πρόοδους πρέπει να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες ε, ώστε το βάρος ε, που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις να μειωθεί για να υπάρξει η δυνατότητα να βελτιωθεί η πρόσβαση ε, των πολιτών και έχουμε μια πραγματικά πολύ αξιοπρόσεκτη προσπάθεια που έχει γίνει στην Πορτογαλία σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε ένα πρόβλημα στόκ πολύ σημαντικό όσον αφορά την, το χρέος των επιχειρήσεων και έχουμε και μια στρατηγική από πλευράς μας για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης επιχειρήσεων. Είναι υποεξέλιξη, αυτή η, ε, έχει δρομολογηθεί αυτή η δράση και τους επόμενους, το επόμενο έτος θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δράση και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα ελπίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ καταρχάς για την επίσκεψή σας. Ακούγοντάς σας κανείς ε, εκπλήσεται ή τουλάχιστον εγώ εκπλήσουμε, διότι έχω την εντύπωση ότι αντιβαίνετε στα όσα είπε ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ, διότι ενώπιόν μας εδώ είπε ότι δεν θα πρέπει να ε, ξαναχρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της Τρόικας. Μήπως διαφωνείτε εσείς με αυτή την πρόταση και δεν ξέρω πώς καταφέρετε να έχετε, να, πώς εξελίχθηκε μάλλον το θέμα της ανεργίας ε, στην ε, Πορτογαλία, αλλά ακούγοντάς σας ε, μάλλον οδηγείτε μένα στην ανεργία, διότι ήμουν εισηγήτρια για το θέμα της δέσμης των 6 μέτρων και ακούγοντάς σας εσάς η οικονομία στην Ευρωζώνη λειτουργεί απόλυτα καλά. Ε, τέλος πάντων, για να σοβαρευτούμε λίγο, Θεωρείτε ότι στα όσα λείπουν από αυτή την οικονομική διακυβέρνηση θα έπρεπε ίσως ε, να έχουμε περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τι άποψη έχετε εσείς για αυτές τις διάφορες εκδοχές που ακούγονται από εδώ και από εκεί και στόχο έχουν να υπάρχει ένα ελάχιστο επίδομα ανεργίας και για να υπάρχει ένα κατώτατο επίπεδο κοινωνικής στήριξης, αλλά για να υπάρχει και μια δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης σε επίπεδο ευρωζώνης. Δεύτερη ερώτηση. Όσον αφορά τις επενδύσεις, ε, σας ετέθησαν αρκετές ερωτήσεις και είπατε για σας ότι η ουσία είναι ε, οι επενδύσεις ε, να ξεκινούν στην Ευρώπη, όχι απαραίτητο από την Πορτογαλία και ότι στην Πορτογαλία τίθεται περισσότερο ζήτημα των ιδιωτικών επενδύσεων. Φαντάζομαι βέβαια ότι η Πορτογαλία θα παρουσιάσει και τα προγράμματά της τα προγράμματα τα οποία θα προταθούν θα είναι προγράμματα τα οποία δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα ή θεωρείτε ότι η Πορτογαλία δεν χρειάζεται αυτό το σχέδιο των επενδύσεων. Τι προσέγγιση έχετε εσεί ω Υπουργό Οικονομικών ε, της Πορτογαλίας ε, για αυτό το σχέδιο των επενδύσεων. Θεωρείτε ότι ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε, ο τρόπο με τον οποίο ε, ε, διαρθρώθηκε μπορεί να αποτελέσει ε, κινητήριο μοχλό της έναρξης των επενδύσεων στην Πορτογαλία που εξετάζω εδώ την ανεργία και το χρέος της Πορτογαλίας εξακολουθεί να είναι λοιπόν μια ευάλωτη χώρα τι αξιολόγηση κάνετε εσείς για το πρόγραμμα αυτό για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευρωβουλευτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πράγματι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σαφώς ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι η ολοκλήρωση, η αρχή, η πορεία και η ολοκλήρωση της Ευρώπης. Θέλουμε όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Ε, ε, απαλήφοντας τις διαφορές και τις ανισότητες και τον κατακαιρματισμό. Έγινε λόγος ήδη για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ε, να μπορέσει ο κατακαιρματισμός στα χρήματα οικονομικά να σταματήσει και η άρση των φραγμών και εμποδίων σαφώς είναι κάτι που θα δώσει δυνατότητες ανοιχτές οικονομίες όπως θέλουμε να είναι η Πορτογαλία και βρισκόμαστε στις παρυφές στην περιφέρεια της Ευρώπης και θέλουμε όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρώπης και ξέρουμε σαφώς ότι η πορεία πρέπει να περάσει από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ίσως δεν κατέστη δυνατό να καταστεί σαφές αυτό που είπα. Έχει ένα πρόγραμμα η, Ευρωπα... Ε, η Πορτογαλία που είναι πολύ καλοδεχούμενο, για να αναζωογονηθεί η, ε, πορτογαλική και η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη. Έχει προγράμματα η Πορτογαλία για να πετύχουν πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο προϋποθέσεων. Πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση επαρκής, πρέπει να υπάρχει μια βάση κεφαλαίου που θα υποστηρίζει την ε, χρέωση και πρέπει να υπάρχει κυρίως εμπιστοσύνη γιατί οι επενδύσεις χρειάζονται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αυτό πρέπει να επιτευχθεί στην Πορτογαλία και αυτό ε, πάλι εξαρτάται από την εξέλιξη των πραγμάτων στη ζώνη ευρώ. Δεν είπαμε ότι δεν θέλει να υποφεληθεί η Πορτογαλία ή δεν θα υποφεληθεί σε σχέση με την μόχλευση των ε, ιδιωτικών επενδύσεων. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα γίνει αυτό. Αλλά επίσης θα υποφεληθεί η Πορτογαλία σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των προγραμμάτων και για την ε, ανάπτυξη όσον αφορά των κυριότερων εταίρων μας και όχι μόνο από τις άμεσα ωφέλη για τη δική μας επικράτεια αλλά και από τις άλλες ε, επενδύσεις που θα φέρουν έμεσα ωφέλη σε μας. Δηλαδή όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θα δώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για τη χώρα μας που γεωγραφικά βρίσκεται στην περιφέρεια της Ευρώπης και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φραγμοί και τα εμπόδια που ακόμα υπάρχουν σταδιακά να μπορέσουν να αρθούν. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συνεχίζει να είναι ευάλωτη η πορτογαλική οικονομία και στην αρχική μου παρέτηση αυτό είπα, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και πρέπει να υπάρχει στένος και συνέχεια προσπάθειας που θα ακολουθηθεί και θα γίνει, ώστε οι βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί να εμβαθυνθούν και να μπορέσουν να εδραστούν καλύτερα ώστε να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει θετικά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Υπουργό ανάμεσά μα Υπουργό Οικονομικών και να υπογραμμίσω ότι είναι ιδιαίτερα ικανή και έχει ιδιαίτερο στένος και είναι ιδιαίτερα νυφάλια και σοβαρή πολιτικά. Το πρόγραμμα προσαρμογών όπως ε, πραγματικά ε, ακολουθήθηκε ήταν ε, μια επιτυχία. Υπάρχουν όμως παράπλευρες απώλειες και αρνητικά στοιχεία παράπλευρα. Απαιτήθηκε τεράστια προσπάθεια των Πορτογάλων, των οικογενειών τους και των επιχειρήσεων. Μετά από αυτό το διάστημα ερωτώ ποια μαθήματα μπορούμε να συναγάγουμε από αυτό το πρόγραμμα. Ποιες συμβουλές μας δίνετε για το μέλλον από όλα αυτά. Ποιες αλλαγές θα προτείνατε. Δηλαδή ποια μαθήματα μπορούμε να αρθρώσουμε και να συναγάγουμε. Και μια ε, παράλληλη ερώτηση. Το αρχικό σχέδιο που είχε συλληφθεί μάλιστα με υπευθυνότητα η συμφωνία του προηγου... της προηγούμενης κυβέρνησης σε σχέση με το πρόγραμμα ε, προσαρμογών. Ήταν καλό και θετικό αυτό όπως είχε αρχικά. Και τώρα για την ε, παγίωση είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα επιτεύγματα. Η ερώτηση όμως είναι πώς ε, θα συνεχιστεί αυτή η καταπολέμηση των απατών και της φοροδιαφυγής και εις φοροδιαφυγής. Υπάρχουν εδώ προβλήματα για τον προϋπολογισμό. Ποια μέτρα είναι εκείνα που θα μπορούσε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Να είναι πιο επιτυχής ε, η καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Απάντηση ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά. Πράγματι το θέμα των προτερημάτων ή μη προτερημάτων του προγράμματος. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν ποτέ να μην ήταν αναγκαίο ένα τέτοιο πρόγραμμα για την Πορτογαλία. Σε αυτή την πτυχή συμφωνώ φυσικά με τον πρόεδρο Γιούγκερ ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχε Τρόικα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάγκη να έρθει Τρόικα στην Πορτογαλία. Δηλαδή οι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να βρεθούν σε κατάσταση ε, χρεοκοπίας ώστε να χρειαστεί Τρόικα υπήρχε, εφόσον υπήρξε αυτή η ανάγκη και αυτό απορρέει από ένα σύνολο ολόκληρο κανονισμών και ε, διατάξεων που περιφρονήθηκαν και αμελήθηκαν κατά το παρελθόν και οδηγηθήκαμε στη χειροκοπία η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ ε, μεγάλη επιβάρυνση αυτό το πρόγραμμα για τη χώρα και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση που ρεαλιστικά θα μπορούσε κανείς να είχε προσεγγίσει ήταν το λιγότερο αρνητικό σενάριο για την Πορτογαλία. Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει καθόλου αυτά τα οποία πρέπει να αναφερθούν για τις θυσίες των Πορτογάλων, θυσίες που υπέστησαν οι Πορτογάλοι πολίτες και που συνεχίζουμε να επιβαρυνόμαστε παρότι η κατάσταση βελτιώθηκε. Όμως αυτές οι αλλαγές είναι εκείνες που έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια απόλυτα μια απόλυτη ρήξη, μια μεγάλη σημαντική καμπή σε σχέση με το παρελθόν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα προγράμματα. Εδώ δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ε, πορτογαλικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στις ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συγκριθούν με ύπαρξη άλλων προγραμμάτων για άλλες χώρες. Κάνουμε λόγο για όριμες ε, ε, σε σχέση με τις οικονομίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Καταστάσεις όπου δεν υπήρχαν μέσα στη διάθεσή μας ώστε με συναλλαγματικές ισοτιμίες ή άλλες, άλλους ελιγμούς να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Έπρεπε λοιπόν εδώ πραγματικά μέσα από μια μακροπρόθεσμη διαδικασία να γίνουν οι προσαρμογές. Και έτσι ουσιαστικά με βάση την πραγματικότητα προχωρήσαμε. Τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε ένα εξωτερικό πλαίσιο που ήταν πολύ λιγότερο ευνοϊκό από εκείνο το οποίο αρχικά είχαμε προβλέψει είχαμε σχεδιάσει με κατάσταση πληθωριστική πολύ χαμηλή σε χαμηλά επίπεδα μια, ας το πω έτσι, πιο δύσκολη κατάσταση οικονομικών συντελεστών και στοιχείων. Σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα τώρα, στόχευε στα τρία κυριότερα προβλήματα την ανάγκη εξυγίανσης ε, των δημοσιονομικών, ανάκαμψης της σταθερότητας της ε, οικονομικής και επανόρθωση των μη ισόρροπων σχέσεων ε, οικονομικών. Υπό αυτό το πρίσμα η λογική του σχεδιασμού αυτού του προγράμματος ήταν σωστή λογική. Μόνο που έπρεπε να είχε γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ πιο εύκολο να το λέει κανείς αυτό τώρα, αφού συνέβη αυτό προηγούμενα. πώ έπρεπε δηλαδή να είχε σχεδιαστεί αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τότε που έγινε. Και πάνω απ' όλα όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι ήταν δυνατόν να επανορθωθούν αυτά μακροπρόθεσμα. Και έχουμε κάποιες ε, ε, εκτιμήσεις που ήταν ιδιαίτερα σκληρές, ε, κάποιες ε, δράσεις και με βάση εκτιμήσεις που ήταν ιδιαίτερα σκληρές. Αλλά καταφέραμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις αγορές. Μία οικονομία που ήδη από πέρσι έχει αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και έχουμε ένα ποσοστό ανεργίας που είναι απαράδεκτα υψηλό, σίγουρα, όμως μειώνεται, μειώνεται σταδιακά με συνέπεια, με συνεκτικότητα. Έχουμε προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όμως οικοδομούμε το μέλλον με βάση πιο στερεές βάσεις, πιο αξιόπιστες βάσεις σε σχέση με τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στο παρελθόν, σε σχέση με την απάτη, τις απάτες και τη φοροδιαφυγή. Έχουμε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και σε σχέση με το 2014 που δεν υπήρξε αύξηση της ε, φορολογήσης αλλά υπήρξε πολύ σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη που ε, συνεισέφερε. Ήταν λοιπόν αποτελεσματική η δράση ε, σε σχέση με τους μηχανισμούς που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μπορούν ακόμα να βελτιωθούν αυτοί οι μηχανισμοί για να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Στο μέτρο που θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, στον μέγιστο βαθμό αυτά τα μέσα και αυτά τα εργαλεία στο πεδίο εφαρμογής θα έχουμε ακόμα την δυνατότητα όταν να αυξηθεί η επιτυχία μας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των, των απατών. Και για το ότι ήταν δυνατόν να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα και που δείχνουν ότι η κατάσταση στην Πορτογαλία βελτιώθηκε πολύ σημαντικά. Σήμερα η Πορτογαλία βρίσκεται μεταξύ των χωρών εκείνων που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχουν το, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα φοροαπατών και φοροδιαφυγής. Πρέπει όμως να δούμε και το θέμα αυτό περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς ένα καλύτερο εναρμονισμό φορολογικό και πρέπει οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στον ανταγωνισμό να αντιμετωπιστούν εφόσον ακόμα συνεχίζουν και υφίστανται και να μπορέσουμε όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα, τη μάστιγα των απατών. Ευχαριστώ. Λούντβινσον, παρακαλώ στη συνέχεια. Eh, Η Πορτογαλία έχει ένα δίκτυ ανεργίας των νέων πάρα πολύ υψηλό. Κάνουμε λόγο για ποσοστά 35 περίπου τα 100. Αν κατανοώ καλά την κατάσταση, αυτή τη στιγμή εσείς εφαρμόζετε μέτρα για να, να προωθήσετε την απασχολησιμότητα των νέων. Και ρωτώ για αυτή την απασχολησιμότητα. Πώς λειτουργήσαν μέχρι σήμερα αυτά τα μέτρα για να προαθεί η απασχόληση σε σχέση με τους νέους. Ποια αποτελέσματα μπορούν να έχουν αυτά τα μέτρα κατά το μέλλον και ποια είναι τα μελλοντικά σε σχέδια και προγράμματα όσον αφορά τους νέους και μια ενεργό πολιτική για την αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρωβουλευτά. Πράγματι, αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχει η Πορτογαλία το υψηλό ποσοστό ανεργία των νέων. Αλλά δεν είναι αποκλειστικό τη Πορτογαλία αυτό το χαρακτηριστικό. Η ανεργία αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα του Πορτογάλου και η ανεργία των νέων είναι τεράστια διασπάθηση δυναμικού. Έχουμε μία γενναία που είναι καλύτερα προετοιμασμένη σήμερα από ότι οι γενναίες του κατά το παρελθόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ακολουθώντας πρότυπα ευρωπαϊκά και προγράμματα της εγγύησης για τους νέους, για την νεότητα για παράδειγμα. Θέσαμε αυτούς τους μηχανισμούς και τους δρομολογήσαμε για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτή τη μάστιγα, την εμβέλεια αυτής της μάστιγας. Και όσον αφορά για παράδειγμα τα μαθήματα κατάρτισης ε, στάζ, υποστήριξη του προγράμματος ε, εγγύησης για τους νέους, δημιουργία μαθημάτων κατάρτισης επαγγελματικής για τους νέους στις επιχειρήσεις και ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων μέχρι τα τέλη του προηγουμένου έτους. 70% των νέων μετά από αυτό το στάζ, μετά από αυτά τα μαθήματα κατάφεραν να βρουν απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που χρειάζονται οι νέοι τις περισσότερες φορές είναι αυτή η πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή, πηγαίνοντας να βρουν εργασία, πρέπει να έχουν κάποια πείρα. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη πείρα ή εμπειρία, είναι ένας φαύλος κύκλος, δεν τους δίνει κανείς δουλειά. Με αυτά τα προγράμματα τα οποία δρομολογήσαμε, κατάφεραν να στεφθούν με επιτυχία και αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν μέχρι πέρυσι, από αυτά 70% των νέων που ολοκλήρωσαν τέτοια μαθήματα μπόρεσαν να βρουν θέση απασχόλησης. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτές τις πολιτικές δρασ, ε, ε, ε, ενεργούς ανάπτυξη, ενεργού ανάπτυξης των, των, της αγοράς εργασίας για τους νέους με τέτοιες δράσεις. Πρέπει να στοιχηματίσουμε επίσης στην επαγγελματική κατάρτιση πιο τεχνικού χαρακτήρα κατάρτισης. Για ιστορικούς λόγους τώρα δεν είναι αυτή η στιγμή να επισέθω σε αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ζητώ συγγνώμη στην Πορτογαλία σταμάτησε η παράδοση της επαγγελματικής κατάρτισης στα σχολεία και δεν πήγαιναν μετά στη συνέχεια οι νέοι στο πανεπιστήμιο και έτσι σε σχέση με την επαγγελματική τους κατάρτιση δεν βρισκόντουσαν στην καλύτερη κατάσταση. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, βέβαια αυτό είχε βαθύτερες ρίζες, υπήρξε μια πιο επαγγελματική μορφή κατάρτιση και εκπαίδευση, δίνοντα δυνατότητα στου νέου, ακόμα και αν δεν είχαν ανώτερε σπουδέ, να αποκτήσουν ένα επάγγελμα και δεξιότητε ώστε να μπορούν να βρουν απασχόληση οι νέοι μας. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε ακόμα να έχουμε ανεργία νέων αρκετά υψηλή σημειώθηκαν μίο μειωτικές τάσεις, τάσεις ε, μείωσης αυτών των ποσοστών. Συνεχίζουμε την πολιτική απασχόλησης, ε, στοιχηματίζουμε στην κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων, ώστε στην αγορά εργασίας να μπορέσουν να ενταχθούν. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την ελαστικότητα και ευληγησία. Το είδαμε αυτό και το επαληθεύσαμε ότι σήμερα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μείωση των ε, προσωρινών ε, συμβολέων απασχόλησης, μερικής απασχόλησης. Έχουμε λοιπόν μια πιο σταθερή θέση των νέων στην εργασία. Πρέπει όμως να πούμε ότι σε αυτό δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια και να πούμε εντάξει το λύσαμε το πρόβλημα. Όχι. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και να συνεχίσουμε με δράσεις ε, από πλευράς της κυβέρνησης και μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Speaker is επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Ε, να σας κάνω ένα κοπλιμέντο όχι για την πολιτική που μας παρουσιάσατε, αλλά και για τις συνέπειες ε, στην Πορτογαλία. Διότι με την αλλαγή της κυβέρνησης είχε τεράστια προβλήματα η χώρα και εσείς με την απαραίτητη επίταση και έμφαση καταφέρατε να αποφύγετε την πτώχευση. Αυτό δεν ήταν εύκολο και απλό για τους εμπλεκομένους, αλλά οι προηγούμενες σοσιαλιστικές αμαρτίες δεν μπορούν να έρθουν μια νυχτή. Η ανταγωνιστικότητα ε, ε, ε, υπέφερε με υπερβολικές ε, ε, μισθολογικές αυξήσεις, για παράδειγμα αυτά ήταν σφάλματα που μείωσαν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη συνολικά. Επίσης θέλω να, θέλω σας συγχαρώ, αλλά και να ρωτήσω κάτι. Αν δείτε το παρελθόν, τα μέτρα της Τρόικας, γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα την επικρίνουν την Τρόικα, ε, συνήθως συμφωνούν με τις προτάσεις της Τρόικα και η Πορτογαλία το έκανε. Αυτά τα μέτρα της Τρόικα λοιπόν και ο θεσμός της Τρόικα, ε, είπε η κυρία ε, Μπερές ότι θέλει να μεταρρυθμίσει την Τρόικα ο Γιούγκαρ, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τα μέτρα της Τρόικα σε τελευταία ανάλυση είχαν νόημα ή θα λέγατε σε τελευταία ανάλυση ότι κάναμε περισσότερα από ό,τι πρότεινε η θα λεγατε σε τελευταια αναλυση οτι καναμε περισσοτερα απο οτι ειναι η τροικα και γι' αυτό τα καταφέραμε. Τέλος, στην Ελλάδα για παράδειγμα, την εμπειρία σας, αλλά και σε άλλες χώρες, ε, στη Λετωνία που είναι εκτός Ευρωζώνης. Θα, θα μπορούσατε στην Ελλάδα να συστήσετε να έχουν έναν αποτελεσματικό, να προσλάβουν έναν αποτελεσματικό Υπουργό Οικονομικών όπως είστε εσείς. Δηλαδή οι μεταρρυθμιστικές ανάγκες φαίνεται να λιμνάζουν στις μεγάλες χώρες και οι μικρές ε, προχώρησαν αποτελεσματικά και γι' αυτό σας αξίζει έπαινος. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα πρόγραμμα προσαρμογής πάντοτε λαμβάνει χώρα σε δύσκολη περίοδο. Πάντα είναι δύσκολο για το λαό. Χρειάζεται πειθαρχία, αυστηρότητα και η προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει με μηδενικό κόστος. Υπάρχουν θυσίες ε, κυρίως όταν πρόκειται για απάλληψη μεγάλων διαρθρωτικών ανισοτήτων. Ε, Προφανώς πλήττεται ο πληθυσμός. Η κυβέρνησή μας προσπάθησε να περιορίσει το κόστος αυτό το κοινωνικό με μια ε, δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι. Και αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια προσαρμογής δεν έπεσε στους ώμους των μικρών, των αδύναμων, αλλά η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα επιβαρύνθηκαν. Ήταν δύσκολα χρόνια όμως αυτά για όλους μας, τρία δύσκολα χρόνια. Και οι θυσίες όμως είχαν νόημα. Τώρα που βλέπουμε τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ναι, είχαν νόημα οι θυσίες μας γιατί ε, πρόοδοι υπάρχουν σε όλους τους τομείς του προγράμματος. Έγιναν μεταρρυθμίσεις, συνεχίζονται και χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον της Πορτογαλίας. Ε, ε, συνομιλήσαμε πάρα πολύ εντατικά με την Τρόικα, μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και με τα επιμέρους θεσμικά όργανα, γιατί εμείς στην αρχή είμαστε σε σχετικά αδύναμη θέση. Ε, τώρα ε, υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και είχαμε μια γνήσια συνεργασία. Δηλαδή ήταν η εταίρη μας η Τρόικα, έτσι τους είδαμε ως παράγοντες αυτής της διαδικασίας και έπρεπε να ε, εφαρμοστεί το, το πρόγραμμα της Τρόικα. Και, μέσα, και επίσης ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία μας έδειξαν και κατανόηση. Και γι' αυτό μεταξύ άλλων είχαμε τα καλά αποτελέσματα. Ξέρω ότι πρέπει να περάσουν και άλλες χώρες από τέτοια προγράμματα. Ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Εκοφίν, πάντοτε αναφέρεται αυτό το θέμα ότι έπρεπε να ζοριστεί πολύ η Ελλάδα και άλλες χώρες. Είναι συλλογική προσπάθεια που πρέπει να την επομιστούμε όλοι και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει επίσης να κάνουν προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται εδώ συλλογική προσπάθεια. Τώρα δίνω το λόγο στον τελευταίο μιλητή γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας και περιμένουν για την ακρόασή μας διακεκριμένοι ομιλητές. Ο κύριος Κώστας Μαυρίδης. Ευχαριστώ, θα είμαι συντομότατος. Κυρία Υπουργέ, πριν από ένα μήνα και λιγότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια έκθεση επέκριναν την Πορτογαλική κυβέρνηση και μεταφράζω εδώ από μια εφημερίδα μπροστά μου. Σε κάποιες περιπτώσεις πολλά από τα θετικά επιτεύγματα αντεστράφησαν. Θέλω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Δεύτερον, δεν θα ρωτήσω για την ανεργία, γιατί μπορεί να τσακωνόμαστε επί ώρες σχετικά με το πόσο μακροπρόθεσμη είναι η μακροπρόθεσμη ανεργία. Άλλη ερώτηση. Όταν μια χώρα βγει από το πρόγραμμα της Τρόικα, υποθέτουμε ότι αυτό θα πρέπει να έχει άμεσο αντίχτυπο στα χαμηλότερα επιτόκια και στον όγκο που μπορεί να δανειστεί για την αναδιάρθρωση η χώρα αυτή, τον όγκο δανεισμού. Ισχύει αυτό για την Πορτογαλία. Τρίτον, υπάρχει κανένα θετικό δίδαγμα για χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα κλπ. Υπάρχει ένα δίδαγμα αποφυγής και ένα δίδαγμα ε, υιοθέτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε μια πρώτη φάση του προγράμματος υπήρχε κριτική, υπήρχαν επικρίσεις προς την κυβέρνησή μας και δεν συμφωνούσαμε πάντοτε σε σχέση με αυτά που είχαμε πετύχει και εν μέρη ισχύει αυτό ότι κάποια θετικά αποτελέσματα ανατράπηκαν, αλλά όλο το πρόγραμμα έχει μεγάλο συμβολικό νόημα. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Και αυτό είναι θετικός, γιατί οι μεταρρυθμίσεις εξετάστηκαν, προσαρμόστηκαν ε, αναλύθηκαν σε βάθος, είδαμε πολύ συγκεκριμένα πώς επηρέασαν την πραγματικότητά μας οι μεταρρυθμίσεις και καμιά φορά υπήρχε στη μεταβατική περίοδο από τη μία φάση στην άλλη κάποιο πρόβλημα κατανόησης, μετάβαση ας πούμε από το πρόγραμμα καθ' αυτό στο μετέπειτα πρόγραμμα, στο διάδοχό του. Ίσως δεν ε, γινόντουσαν όλα εκεί σωστά κατά τη μεταβατική περίοδο. Αλλά δεν πιστεύομαι ότι η κρίση είναι αρνητική συνολικά. Συνολικά το πρόγραμμα πήγε καλά. Ε, έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις. Τώρα έχουμε δύο μεγάλες αφρολογικές μεταρρυθμίσεις. Ε, θα δημιουργηθεί ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο στον προϋπολογισμό και στον ενεργειακό τομέα έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα. Κανένα τομέα δεν αφήνουμε απ' έξω. Παντού προσπαθούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι καμιά φορά αυτά δεν γίνονται τόσο καλά ε, κατανοητά. Ε, δεν, δεν υπάρχει σωστή αντίληψη για το τι κάναμε. Η μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια δεν ε, χαλάρωσε, αντίθετα. Ε, τώρα, όταν μια χώρα βγαίνει από το πρόγραμμα, τι γίνεται με τα επιτόκια. Εμείς έχουμε ιστορικά χαμηλά επιτόκια αυτή τη στιγμή και αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τα βράχη και μέσο πρόθεσμα ομόλογα που εκδίδει το δημόσιο. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή έχουμε κάνει κάποια σχέδια για το 2015 και το 2016, ώστε οι επενδυτές να, αποκτή, να έχουν κάποια ασφάλεια, να νιώθουν κάποια ασφάλεια, να είναι εξασφαλισμένοι τέλος πάντων. Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή τη διαδικασία του χρέους σωστά. Αυτό που προσφέρει η αγορά είναι καλό, είναι θετικό. Αντιδρά θετικά η αγορά, αντιδρούν θετικά οι αγορές. Αυτό άρχισε να φαίνεται και πριν από το τέλος του προγράμματος, αυτή η νέα κατάσταση που διαμορφωνόταν. Αλλά τώρα υπάρχει διαφάνεια στις αγορές, μπορούμε πραγματικά να το πούμε αυτό, οι επενδυτές έχουν εμπιστοσύνη στην πορτογαλική οικονομία και όπως σας είπα τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και αυτό σημαίνει προφανώς ότι η κατάστασή μας θα βελτιωθεί στο μέλλον. Με περισσότερη σταθεροποίηση, μεγαλύτερη σταθερότητα και στη ζώνη του ευρώ αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την συμβολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι αυτή την αξιοπιστία στις αγορές να την ξανακερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, κυρία Υπουργέ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η επαφή, αυτός ο οικονομικός διάλογος. Εκφράζω επίσης την επιθυμία στο μέλλον η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να προσπαθήσουμε να αποφύγει το γεγονός, να αποφευθεί το γεγονός ότι ανήκουμε ή μεν σε μία ή άλλη ή δε σε κάποια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να προσεγγίζουμε καταστάσεις αμφωτέρωθεν, όπως το είδαμε και σήμερα το πρωί. Και ελπίζω ότι στο μέλλον θα προσπαθήσουμε πιο ενωμένοι να προσπαθήσουμε να δράσουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Να είμαστε το δυνατόν πιο αντικειμενικοί στις συζητήσεις και αξιολογήσεις μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ κυρία Υπουργέ Οικονομικών της Πορτογαλίας για το ότι ήρθατε εδώ ενώπιόν μας. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Δημόσια κρύωση, ακρόαση σχετικά με τη διατροτική μεταρρύθμιση των τραπεζών. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, ομιλητές μας, 7 τον αριθμό για τη σημερινή ακρόαση, για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, για τη δημοσιονομική σταθερότητα και επίσης η ακρόαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τις εργασίες μας ε, ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013 σε μία έκθεση ίδιας πρωτοφουλίας ε, εξέτασε διαρθρωτικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι απαραίτητα για να συμπληρώσουν άλλε μεταρρυθμίσει για την εποπτεία, την εξυγίανση και τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει για να αντιμετωπίσουμε το too big to fail, too big to save και να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προβλήματα. Και φυσικά αυτό ε, συνάδει και με τα συμπεράσματα τη έκθεση, τη ομάδα υψηλού επίπεδου, στην οποία προείδρευε ο πρόεδρος Λίκανεν, ο οποίος είναι εδώ σήμερα και τον οποίο καλωσορίζω θερμά. Και τώρα φυσικά μετά από δύο χρόνια από το ψήφισμά μας, ε, ε, δύο περίπου χρόνια από την έκθεση Λίκανεν και λόγω και της συγκεκριμένη πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και της θέσης σε ισχύ των νέων διατάξεων για την εποπτεία, και τη μελλοντική θέση σε ισχύ της, ε, των διατάξεων για το bail-in, για τη διάσωση με ιδιοσπόρους και τις κεφαλακές απαιτήσει και λόγω και της πολύ μεγάλης ε, διάστασης ε, των στοιχείων ενεργητικού του των τραπεζών, είναι απόλυτα επίκυρη η συζήτηση με εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά της υποχρεωτικής, του υποχρεωτικού διαχωρισμού των διαφόρων δραστηριοτήτων, καθώς και τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις που έχουμε για τις διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις. Είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση αυτή και είμαι βέβαιος ότι η ακρόαση αυτή θα μας ε, ε, προσφέρει και πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία για την εξέτασή μας. Ε, αποφασίσαμε να ε, διαρθρώσουμε την ακρόαση σε δύο συνεδρίες. Η πρώτη έχει τίτλο ε, «Είναι οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες εγγενώς επικίνδυνες» και η δεύτερη «Ποιες είναι οι συνέπειες των διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων για τη διαφορετική μεταρρύθμιση». Θα δώσουμε 7-8 λεπτά στους κάθε, στον κάθε ομιλητή για να κάνουν κάποιες αρχικές παρατηρήσεις. Σας παρακαλώ τηρήστε αυτό το χρονοδιάγραμμα και να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα προκειμένου να γίνεστε κατανοητοί μετά από τις ε, παρατηρήσεις από ε, το πάνελ θα δώσουμε και το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Πρώτος ομιλητής, ε, δεν χρειάζεται καμία σύσταση, ο Έρκη ο οποίος ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος από το 1995 μέχρι το 2004 και τώρα υπηρετεί τη δεύτερη θητεία του ως ε, διοικητής της Τράπεζας της Φιλανδίας και σήμερα ε, είναι εδώ ως πρόεδρος ε, της ομάδας υψηλού επίπεδου για την μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Λίκανεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανάλυση τη ομάδα υψηλού επίπεδου για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από δύο χρόνια αποκάλυψε ότι έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα ε, στα διάφορα τραπεζικά μοντέλα, αλλά κυρίω ε, σε πολύ περίπλοκα μέσα με δραστηριότητες οι οποίες ε, πολύ ε, γρήγορα κλιμακώνονται. Προτάθηκε λοιπόν μια μεταρρύθμιση που θα μειώσει τα κίνητρα για πολύ ε, υπερβολικούς κινδύνους, ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες των τραπεζών. Και καταλήξαμε στο ε, συμπέρασμα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, ε, οι τράπεζες και να οδηγηθούν ε, να αυξήσουν τη μόχληση, να μεγαλώσουν και να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους χωρίς να υπάρχουν ταυτόχρονα οι κυβερνητικές εγγυήσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν. Επομένως το βασικό ερώτημα για αυτό το πρόβλημα του big to fail είναι αν έχουμε κάνει αρκετά ώστε να διαγραφεί αυτό το πρόβλημα. Ε, στις συζητήσεις μας καθορίσαμε δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος ε, προτείνει ε, οι εύρωστες κεφαλαϊκές απαλλητήσεις, οι οποίες δεν βασίζονται σε περίπλοκα μοντέλα, να επιβάλλονται για τις εμπορικές δραστηριότητες. Και επιπλέον οι εμπορικές δραστηριότητες θα πρέπει να διαχωρίζονται αν μια τράπεζα δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης δεν είναι αξιόπιστα. Στο δεύτερο δρόμο θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των σημαντικών εμπορικών δραστηριοτήτων από τις ε, ε, ε λιανικές τραπεζικές ε, δραστηριότητες. Επιπλέον κεφαλαϊκές απαιτήσεις δεν θα επιβάλλονται σε αυτή την περίπτωση, αλλά ο διαχωρισμός θα πρέπει να πληρεί τις συγκεκριμένε ε, κεφαλαϊκές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας. Μετά από συζήτηση καθορίσαμε ότι ε, ε, ε, το επίπεδο της εμπορικής δραστηριότητας υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώτατο όριο. Θα ήθελα λοιπόν να επανεξετάσω αυτά τα βασικά ερωτήματα σήμερα με τέσσερις διαφορετικές πτυχές. Καταρχάς, η επίλυση των μεγαλύτερων και πιο έντονης δραστηριότητας εμπορικής τραπεζών είναι αξιόπιστη ακόμα και σε περίπτωση πολύ μεγάλων πιέσεων η οδηγία για την ε, ε, εξυγίανση και την αναβάθμιση των τραπεζών ε, μας δίνει πολύ σημαντικά εργαλεία για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ε, τράπεζες οι οποίες κινδυνεύουν να πτωχεύσουν με πολύ καλό τρόπο και χωρίς να επιβάλλουμε επιπλέον επιβάρυνση στους Ευρωπαίους φορολογημένους. Επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι μεγαλύτερες και οι τράπεζες οι οποίες έχουν μεγαλύτερες εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να εξυγιανθούν γρήγορα εν μέσω συστημικής κρίσης. Εάν ε, η δομή ε, μιας τράπεζας έχει απλουστευτεί εκ των προτέρων, θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλλουμε μέτρα εξυγίανσης, ακόμα και όταν υπάρχουν πολύ σοβαρές πιέσεις. Δεύτερον, μπορούμε να περιορίσουμε τη διάχυση των ωφελών από το σύστημα εγγυήσεων των καταθέσεων και οποιαδήποτε σε ε, κυβερνητικέ εγγυήσει για κάποιε εμπορικέ δραστηριότητε των τραπεζών. Ε, το να είναι οι εμπορικές δραστηριότητες αξιόπιστη επιλογή θα μειώσει ουσιαστικά την εγγύηση για τις τράπεζες, αλλά ε, μπορεί να εποφοληθούν οι καταθέσεις από μια συγκεκριμένη εγγύηση των τραπεζών ως βασική δραστηριότητα, ε, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολύ ισχυρές πιέσεις χωρίς διαχωρισμό ε, και άλλες ε, τραπεζικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να επιφαληθούν από αυτή την ε, υπόλοιπη εγγύηση των τραπεζών και έτσι θα μπορούμε να έχουμε ένα πεδίο εφαρμογή που ίσως θα είναι ευρύτερο από όσο θα έπρεπε και μπορεί να δημιουργεί και περισσότερες θευλώσεις οι δραστηριότητες σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να υποσκάψουν ε, την ε, ε, δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτό ισχύει κυρίως όταν υπάρχει υπερβολική ανάπτυξη και αναλαμβάνονται πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Και αυτό ισχύει κυρίως όταν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό άειλων στοιχείων αποθεματικού και έτσι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε διάκριση δραστηριοτήτων που είναι ε, για τη δημιουργία της αγοράς από τις ε, ε, εμπορικές δραστηριότητες ιδιοκτησίας. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει κατάλληλη προστασία από πιθανούς υπερβολικούς κινδύνους στην εμπορική δραστηριότητα. Ε, οι κεφαλαϊκέ αποτίσεις θα πρέπει ε, να αντανακλούν πλήρω του τους κινδύνους που αναλαμβάνονται. Κυρίως οι κεφαλαιακές αποτίσεις έχουν τροποποιηθεί ώστε να αντανακλούν καλύτερα τον κίνδυνο των εμπορικών δραστηριοτήτων, της τυκλοποίησης και της έκθεσης των τραπεζών στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Επιτροπής της Βασιλείας για την ε, θεμελιώδη ε, αναθεώρηση του εμπορικού κώδικα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού υπάρχουν ε, αποθεματικά ασφαλείας ε, στα οποία είναι δύσκολο να έχουμε μοντέλα για τους κινδύνους. Και επιπλέον ένα συνδυασμός δραστηριοτήτων υψηλών κεφαλαικών απαιτήσεων ε, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κεφαλαίου που σπανίως θα χρειάζεται για να καλύψουν τις μεγάλες απώλειες. Τέταρτο ερώτημα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι απλές προς παρακολούθηση, εποπτεία και διαχείριση ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματική επιθαρχία και τον ηγετικό ρόλο των αγορών. Τα κίνητρα για τους ε, ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των τραπεζών αυξάνονται μέσω της οδηγίας για την εξυγίαση την αναβάθμιση των τραπεζών και του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις τράπεζες ε, για τα επιχειρηματικά τους μοντέλα εάν δεν υπάρχει ένα ε, υφέρπο σύστημα διακυβέρνησης. Ο διαχωρισμός επίσης για τους νέους επόπτες θα κάνει πιο εύκολα διαχειρίσιμα τα νέα καθήκοντα. Και αυτό ε, ε δημιουργεί τον κίνδυνο μεταφορά στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα και μπορεί φυσικά να υπάρχει και πρόβλημα για την κατάλληλη εποπτεία. Τέλος, οι διαρθρωτικές τράπεζες αν έχουν γίνει επαρκώς απλές μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Πιστεύω ότι ε, η περισσότερη μείωση στην περιπλοκότητα μέσω του διαχωρισμού χρειάζεται προκειμένου να διευκολύνουμε την διαχείριση και την αποτελεσματική εφαρμογή των κινήτρων αφενός για τις τράπεζες καταθέσεων και αφετέρου για τις εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι θα μειωθεί το μείγμα, την ανάμειξη δύο πολύ διαφορετικών νοοτροπιών, μία πιο βραχυπρόθεσμη και μία πιο μακροπρόθεσμη. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να, θέσω, να απαντήσω μάλλον το ερώτημα το οποίο ετέθη. Ε, διότι η μεταρρύθμιση μέχρι τώρα μας έχει οδηγήσει μεν ε, σε πολύ μεγάλο δρόμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος του too big to fail, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, δεν έχουμε βρει την ηθάκη. Είναι λοιπόν ε, ε, ακόμα, δεν είναι παρκώς ισότιμη η ανταγωνισμού και οι μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να <coughs> μεταρρυθμιστούν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίκα. Και ο δεύτερος αγορητής πολύ γνωστός. ο καθηγητής Charles Goodhart, επίτιμος καθηγητής ε, τραπεζικών ε, στο London School of Economics. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου έζησα τρεις τραπεζικές κρίσεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 74, 75, 90, 91, 2008, 2009. Όλες αυτές οι κρίσεις ε, είχαν τα αίτια τους ε, σε δάνεια τα οποία δεν ήταν αξιόπιστα. Ιδίως ε, κιόλας και στο τομέα των ακινήτων και εκτός και εντός Ηνωμένου Βασιλείου. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία και στη ΣΥΠΑ επίσης. Όλες αυτές οι κρίσεις ήταν 17 έτη απήχαν μεταξύ τους. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επόμενη κρίση θα ήταν το 2025 αν υπολογίζαμε αυτό με βάση τη σημερινή ημερομηνία. Αυτά όμως ε, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν ε, γίνει αρκετά σε σχέση με την αντιμετώπιση των τροτών ε, όσον αφορά το τραπεζικό μας θέμα. τουλάχιστον όχι στον τομέα τον διαθωτικό. Όσον αφορά την πιστοληπτική δυνατότητα των τραπεζών για την υποστήριξη της ανάπτυξης, με τις κυριότερες αναλύσεις βλέπουμε ότι τα ενυπόθεκα δάνεια, η ε, στέγαση είναι εκείνη που πολλές φορές ε, οδηγεί στην ε, επέκταση των δανείων. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτή η αύξηση, αυτή η ανάπτυξη οδήγησε στην ανάπτυξη μεγαλύτερη από ότι η ανάπτυξη των καταθέσεων. Και όταν βλέπουμε ότι η πιστοληπτική διεύρυνση σε σχέση με τις καταθέσεις ε, ε, το ένα σκέλος απέχει από το άλλο, ε, δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με τους επενδυτές που δεν έχουν ασφαλιστεί επαρκώς και δεν γνωρίζουν τους κινδύνους. Ακόμα και όταν υπάρχουν κειμενόμενα τέτοια δάνεια, ο κίνδυνος ελοχεύει. Η όλο και αυξημένη αυτή δυσαναλογία όσον αφορά την δανειά δανειοδότηση έχει πραγματικά οξύνει την ε, κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά συστήματα. Έγινε μια προσπάθεια ε, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, ένα πλαίσιο ασφαλείας. Οι τράπεζες επιτάχυναν την κρίση στις περισσότερες περιπτώσεις ε, όπου ήταν σχετικά μικρές λιανικών πράξεων τραπεζικά ιδρύματα όπως η Anglo-Irish ε, Northern rock ε, Κάχασα ε, στην Ισπανία και πολλά παραδείγματα στη ΣΥΠΑ και αλλού. Και η, ο πόθος για ανάπτυξη, η τάση για την ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε αυτές τις τράπεζες. Η IBS είναι ένα τέτοιο θλιβερό παράδειγμα με πολύ μεγάλους κινδύνους, με μεγάλη εμβέλεια. Και βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερη, ιδιαίτερα ε, ύποπτες ε, οι δράσεις της ανάπτυξης, ε, οι πράξεις στα παράγωγα για παράδειγμα, οι συναλλαγές με τα παράγωγα ήταν πράξεις που συνεισέφεραν σημαντικά στην δημιουργία της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και όπως θα γνωρίζετε ε, τα παράγωγα στην Lehman Brothers δημιουργούσαν κέρδη. Όταν δημιουργήθηκαν όμως τα προβλήματα, είχαμε τα προβλήματα στον τομέα των στεγαστικών δανείων. Πρέπει να δούμε ότι ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες πολυμορφοποίησης, πολυσχηδούς διαμόρφωσης των κινδύνων. Και πραγματικά είναι τραγωδία ότι οι μεγαλύτερες κρίσεις αυτές δεν οδήγησαν σε μια εκβάθρον επανεξέταση των μηχανισμών στεγαστικών δανείων. Για παράδειγμα, το The House of Death, Death θα ήταν ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Και βλέπουμε το, τα προβλήματα τα οποία υφίστανται όσον αφορά τις επενδυτικές τράπεζες. Και βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα όσον αφορά την ίδια την αξιοπιστία των τραπεζών και δευτερογενώς ε, και στην ε, χρηματοοικονομική κρίση. Και όλα τα σχόλια που γίνονται είναι σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες τους. Όμως στην πρακτική εφαρμογή οι επενδυτικές δραστηριότητες investive, banking, αυτό το οποίο κάνει είναι διευκολύνονται εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ή να ε, προχωρήσουν σε συναλλαγές με τέτοιου είδους δάνεια. Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι καλύτερη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προβλέπεται ένας πολύ μεγαλύτερος ρόλος ε, για τις επενδυτικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο ευρωπαϊκών τραπεζών ε, εκτός ε, αν θελήσουμε να απεμπολίσουμε αυτόν τον ρόλο και τον εγκαταλείψουμε στους, στις τράπεζες των ΙΠΑ το να προσπαθήσει κανείς ε, να οδηγήσει τις τράπεζες ε, στο να μπορέσουν ε, να μειώσουν το ρόλο τους ως διευκολυντών των συναλλαγών δεν είναι η σωστή λύση. Και μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι η δυνατότητα της δράσης αυτών των τραπεζών θα έχει πάντα σημείο αναφοράς τις συναλλαγές σε ιδιοκτησίες ή ακίνητα όπως για παράδειγμα αναφέρεται και στην αρμόδια έκθεση που δεν καλύπτει πλήρως ε, τις ε, λιανικές, τις συναλλαγές λιανικής από απώλειες ενώ υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για το αντίστροφο. Μια και υπό το ενιαίο σημείο εισόδου οι ε, εταιρείε όσον αφορά το αποθεματικό τους θα μπορούσαν να διαβρωθούν. Είναι γεγονός ότι όλες οι ανεπτυγμένες χώρες σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και τον είπα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζικών συναλλαγών γίνεται από ένα μικρό αριθμό ε, μεγάλων τραπεζών. Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό, αλλά μάλλον θα οφείλεται και στο ρυθμιστικό πλαίσιο και για ε, ε, την αρχή too big to fail πάλι δίνεται η δυνατότητα δανειοληπτικής ε, δράσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει η δυνατότητα αλλαγών ε, και οποιαδήποτε μέτρα θα αποδυνάμωναν τις ευρωπαϊκές τράπεζες ακριβώς τη στιγμή που θα τις χρειαζόμαστε περισσότερο θα έχει σαν συνέπεια να υπάρξουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και Ακούσαμε μια διαφορετική άποψη σε σχέση με την πηγή των ε, χρηματοοικονομικών ε, ασταθειών, την ανάγκη ε, πολυμορφοποίησης και περνάμε στον επόμενο αγορητή για να ακούσουμε τις δικές του απόψεις. Μάρτιν Χέρβικ, καθηγητής που τιμήθηκε πολλαπλά πρόσφατα 2012 το έπαθρο Max Planck για την έρευνα για τις ε, διεθνείς ε, ε, διατάξεις ρύθμισης του τραπεζικού τομέα και είναι μέλος του European Systemic Board. Παρακαλώ έχετε τον λόγο να μας εκθέσετε τις απόψεις σας. Μεγάλες τράπεζες έχουν εγγενείς κινδύνους. Η απάντηση είναι σίγουρα, χωρίς αμφιβολίες, ναι. Και έτσι και οι μικρές εξειδικευμένες τράπεζες εξίσου και εκείνες. Είναι επικίνδυνες οι τραπεζικές συναλλαγές και το κόστος δεν είναι το μέγεθος του κινδύνου, αλλά αν είναι μη ενδεδειγμένοι οι κίνδυνοι, επειδή μπορεί να ελοχεύουν εκεί όπου δεν αναμένονται ή επειδή ε, προέρχονται από όλους τους τομείς. Ε, υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί αυτό το πλαίσιο αν υπάρχουν ε, επαρκή κεφάλαια το αφήνω αυτό το σημείο και θα επανέλθω υστερότερα. Θα κάνω λόγο για τις διαθροτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες. Προτάσεις για διαθροτικές αλλαγές εμπνέονται από την αρχή ότι αυτό θα έδινε προστασία στο χρηματοοικονομικό τραπεζικό σύστημα και στους φορολογουμένους. Πρέπει να δούμε όμως μια συνεκτική επεξήγηση για αυτό το επιχείρημα. Μια πιστική ε, ε, απόδειξη Κάποιες από αυτές τις προσπάθειες εμπνέονται από κάποια νοσταλγική τάση. Ωστόσο αυτή η νοσταλγία δεν είναι η πιο εύθετη προσπάθεια. Κατά το παρελθόν μέχρι το 1970 ήταν ε, σχετικά ασφαλές ε, το χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεν υπήρχαν ε, μεγάλοι κίνδυνοι, τα επιτόκια ήταν σταθερά από το 70 όμως και εφ' εξής, υπήρχαν κίνδυνοι επιτοκίων που άρχισαν να αναφύονται και ισοτιμιών και μεγάλος ανταγωνισμός ε, και το σύστημα κατέστη μη ασφαλές και ήταν πλέον υπεύθυνο στη συνέχεια για την μείζωνα ε, κρίση των ε, τραπεζών καταθέσεων που οδήγησε στην εξειδίκευση των τραπεζών και στην ιστερότερη τραπεζική κρίση που συνέβη το 1990. Πάντα πάλι επειδή ήταν υπερβολικά εξειδικευμένα αυτή τη φορά αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αυταπάτες. Πρώτον, οι εμπορικές δραστηριότητες είναι επικίνδυνες. Η κρίση του 1990 οφειλόταν στα ε, στεγαστικά δάνεια και στα δάνεια ε, απόκτησης ε, πρώτης κατοικίας. Και όσον αφορά τους πιστοτικούς κινδύνους, έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα, ε, μέρος των επικίνδυνων συναλλαγών από ό,τι κατά το παρελθόν. Μια άλλη αυταπάτη, η προστασία των καταθετών και τα συστήματα ε, κάλυψης των καταθέσεών τους. Δεν είναι μόνοι λόγοι ανησυχίας. Οι υποδομές ε, ήταν ένα μείζον πρόβλημα όταν εξαφανίστηκαν οι Lehman Brothers ε, σε σχέση με τις αγορές, την αγορά παραγόγων οι χρηματοοικονομικές αγορές ε, καθώς επίσης και οι ε, δανειοληπτικές δραστηριότητες. Η μείζον επίπτωση των Lehman Brothers στο χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν το ντόμινο, η επίπτωση ντόμινο που είχε σε σχέση με τους ε, πελάτες των χρηματοοικονομικών αυτών ιδρυμάτων που ε, κατέστρεψε ουσιαστικά τον ε, χρηματοοικονομικό ιστό. Ήταν μια επενδυτική τράπεζα η Lehman Brothers το να ε, γίνει κάποια, κάποιος διαχωρισμός δεν σημαίνει ότι επαρκεί και μπορούν να συνεχίσουν όπως πριν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πρώτον η διαχείριση, η διακυβέρνηση. Πώς ε, μπορούν τα κονδύλια, τα ποσά τα οποία ε, βρίσκουν διάβλους και έχουμε την δυνατότητα να περάσουν τέτοιου είδους χρήματα μέσω των ε, Lehman Brothers ε, παρεκκλίνοντας από τον αρχικό τους ε, στόχο που δεν είναι ακριβώς μια ιστορία επιτυχίας. Καθώς επίσης και να δούμε σε σχέση με τις ασφάλειες ενυπόθηκων δανείων πάλι μια ιστορία που δεν στέφθηκε με καμία επιτυχία. Επίσης όσον αφορά επενδυτές και καταθέτες σε γερμανικές τράπεζες, στις Landesbanken των γερμανικών κρατηδίων διοργανώνοντας ένα πλαίσιο εγγυήσεων και ένα ολόκληρο ιστό ε, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ούτε και αυτή είναι μια ιστορία επιτυχίας. Οι επενδύσεις στις Landesbanken βρισκόντουσαν κάτω από τα κατόφλια της προ, ε, νομοθεσίας. Η συμπεριφορά τους λοιπόν θέτει ένα μεγάλο πρόβλημα. Προβλήματα επίσης όσον αφορά την προστασία ε, επενδυτών. Ποια προϊόντα αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και με τις ακροάσεις ε, που έγιναν η πρόσβαση που υπήρχε εμπορικών τραπεζών σε σχέση με επενδυτές ε, εταιρείες που διαμεσολαβούσαν σε σχέση με τους Lehman Brothers. Πάλι ιστορία που δεν στέφτηκε με καμία επιτυχία και η ε, δημιουργία πλεονασματικών ε, ε, δυνατοτήτων κεφαλαιακά επεκτείνεται σε κάτι που θα ήθελα να αποκαλέσω προστασία επαγγελματιών επενδυτών. Είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη κάποιες αρχές προστασίας όταν τα προϊόντα είναι τοξικά και όταν τα χαρτοφυλάκια τα οποία προσπαθούμε να διασφαλίσουμε έχουν βαθμό ανεξαρτησίας στις δραστηριότητές τους. Οι προτάσεις ε, όσον αφορά περιορισμό δραστηριοτήτων καταθετών ε, καθορίζονται υπό τους όρους ποιος μπορεί να επενδύσει και πώς. Όχι όμως με το τι επενδύεται. Τι γίνεται λοιπόν με την εξαγορά τοξικών προϊόντων όσον αφορά ε, τραπεζικές δραστηριότητες, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες επενδυτικού χαρακτήρα. Μετά, ο μολυσματικός χαρακτήρας ε, που μπορεί να έχει συστημικό χαρακτήρα κατά την κρίση των πρώτων ετών 1990 χρησιμοποιούσαν κέρδη από τα α, παράγωγα για να αντισταθμιστούν απώλειες όσον αφορά τις, α, τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ πάλι τίθεται πρόβλημα. Θα έπρεπε να σκεφτούμε διαχωρισμό δραστηριοτήτων σαν μια δυνατότητα ε, πολυμορφοποίησης κινδύνων. Αυτό εξαρτάται από την συνολική αντιμετώπιση κινδύνων και την ε, δυνατότητα μικρότερου όμως εδώ ελέγχου για το τι συμβαίνει. Επίσης ε, συμβάσεις ε, που συνεπάγονται κινδύνους. Δηλαδή πιθανώς μπορεί να υπάρξει ενδυνάμει μεγαλύτερη επίπτωση ντόμινο αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Ταυτόχρονα το δίκτυο αυτών των ε, συμβάσεων μπορεί να είναι πολύ λιγότερο διαφανές από ότι ε, αν είχε κανείς μία μεγάλη ε, παγκοσμιοποιημένη τράπεζα. Όλα αυτά δεν έχουν πλήρως συζητηθεί και αναλυθεί. Δεν γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις. Αλλά αυτές είναι τουλάχιστον κάποιες από τις ερωτήσεις που πρέπει να διατυπωθούν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα τα μέλη θα κάνουν ερωτήσεις στους ομιλητές μας. Ο εισηγητής ε, και οι σκιώδεις θα έχουν δύο λεπτά ο καθένας για ερωτήσεις και θα απευθύνουν συγκεκριμένο ερώτημα σε συγκεκριμένο ομιλητή. Και ο ομιλητής θα έχει τρία λεπτά για την απάντηση. Ο εισηγητής, ο κύριος Κούνερ Χόκμαρ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, για τις ε, παρουσιάσεις αυτές. Όλοι οι προσκεκλημένοι μας ανέλησαν το θέμα των τραπεζών γενικών εργασιών ε, και τον κίνδυνο που ενέχουν, αν είναι μεγαλύτερος. Έχετε σκεφτεί πώς ε, ε, θα είναι οι τράπεζες γενικών εργασιών προς πιο εξειδικευμένες. Θα είναι ας πούμε όταν έγινε μια ανάλυση το 2010 είπαν ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερο σε επενδυτικές ή σε ε, λιανική τραπεζική. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας και ποιο συμπέρασμα θα έβγαινε αν προχωρούσαμε σε διαχωρισμό των τραπεζών γενικών εργασιών. Θα σήμαινε αυτό δηλαδή ότι θα έχουμε πιο πολλές εξειδικευμένες που θα λάμβαναν μεγαλύτερο ρίσκο προς διάφορες κατευθύνσεις και τι θα γίνει με την επενδυτική τραπεζική, επενδυτικές τράπεζες, τράπεζες επενδύσεων. Ε, αν λένε μερικοί ότι αν η τράπεζα εργασιών δεν κάνει ε, επενδυτική τραπεζική, τότε θα έμεναν λίγες που θα ε, προχωρούσαν σε ε, επενδύσεις. Αυτό πώς το βλέπετε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής. Ευχαριστώ. Ποιος θα απαντήσει πρώτος, ο κύριος Λίκανεν. Παρακαλώ. Εμείς ε, στην ε, έκθεση είδαμε πολλά επιχειρηματικά μοντέλα και εξετάσαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν ε, θα λέγαμε ότι ένα μοντέλο, δεν λέγαμε ότι ένα μοντέλο είναι συγκεκριμένα ασφαλές ή ιδιαίτερα ανασφαλές. Επίσης, δεν προτείνουμε να διασπάσουμε τις τράπεζες. Αυτό που προτείνουμε είναι ότι αν ε, ξεπεραστεί ένα κατόφλι, τότε μπορεί να υπάρξει κίνδυνο σταθερότητας και τότε οι εμπορικές δραστηριότητες θα πρέπει να διαχωριστούν παραμένοντας το ίδιο κοντσέρν, αλλά ε, θα πρέπει η κεφαλοποίηση να γίνεται διαφορετικά. Σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες, η Βασιλεία ισχύει για όλους ε, και ε, η έκθεση στο ρίσκο δηλαδή πρέπει να έχει συγκεκριμένα όρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παραμείνουν στο πλαίσιο των ίδιων τραπεζών γενικών εργασιών, χωρίς να διαχωριστούν. Μπορεί να υπάρχει αντίκτυπος όμως, γιατί αν κάποια κόστη αυτών των, αυτε, μάλλον αυτές οι δραστηριότητες ε, που στηρίζονται από εγγυήσεις εκεί μπορεί να ε, γίνουν και αξιολογήσεις αντίκτυπου διαφορετικές. Η κλίμακα των επενδυτικών δραστηριοτήτων θα εξαρτηθούν πολύ από την εξέλιξη της κεφαλαιακής ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, η ε, κεφαλαία μεγαλώσει στην Ευρώπη, τότε οι επενδυτικές τράπεζες ε, θα πρέπει να αυξηθούν ανάλογα. Και υπάρχει ένα όριο. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει η Ένωση. Αυτό θα είναι το ε, όριο. Και σίγουρα συμφωνώ με τον συνάδελφο, τον καθηγητή Χέλβικ, ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι και ήταν μια διακυβέρνηση. Αλλά όσο εξειδικεύεται κανείς, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η εξειδίκευση αυτή ε, συγκεκριμένες δυσκολίες. Και εγώ να προσθέσω δεν νομίζω ότι οι εξειδικευμένε τράπεζες αφεαυτές είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι εξειδικευμένε τράπεζες επενδύσεων είχαν επιτυχία εδώ και δεκαετίε. Μάλλον τα, οι τράπεζες καταθέσεων αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα. Αλλά υπάρχει μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσατε και αυτό επηρεάζει όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λέξη κλειδί είναι ο ανταγωνισμός. Τα τελευταίες τρεις-τέσσερις δεκαετίες είδαμε μεγάλη αύξηση στην ένταση του ανταγωνισμού, ε, πολλές φορές ε, ε, με σκιώδεις τράπεζες ή μέσα από την ανάπτυξη των τραπεζών γενικών εργασιών, αλλά σίγουρα η ικανότητα των τραπεζών ε, έχει διαβρωθεί. Οπότε ε, υπάρχει σε όλες ε, η πιθανότητα κινδύνου. Ο κύριος Γιάκοπ Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τρεις διακεκριμένους ειδικού που έχουν μια, ένα κοινό γνώρισμα, διάβασα καλά τις ε, Εργασία σας. Το κοινό είναι ότι πιστεύετε ότι το πρόβλημα του big to fail δεν έχει ακόμα επιληθεί. Υπάρχουν πολλοί παρευρισκόμενοι και στα πίσω έδρανα κυρίως που λένε ότι εμείς έχουμε ε, κεφάλαιο για διάσωση με ίδια μέσα που θα έλυνε το πρόβλημα. Και ο καθηγητής Χέλβικ και ο καθηγητής Γκούτχαρτ έχουν δημοσιεύσει εργασίες. Ο καθηγητής Γκούτχαρτ μάλιστα πρόσφατα το καλοκαίρι και είπε ότι το κεφάλαιο Μπέιλιν μπορεί να μην είναι το τέλειο υποκατάστατο για άλλα κεφάλαια, όπως το πραγματικό, όπως θα έλεγε ο καθηγητής Χέλβικ, ή το, τα κεφάλαια από τους φορολογουμένους για τη διάσωση των τραπεζών αν ε, έχουμε ε, τέτοιο κεφάλαιο για Μπέιλιν μπορεί να μην ε, ε, δημιουργήσει συστημικό πρόβλημα, αλλά διαρωτώ με και αυτή είναι η ερώτησή μου, αν τα living wills που είναι επίσης προσωρινές ρυθμίσεις είναι καλά υποκατάστατα για διορθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Και για να το αναδείξω αυτό θέλω να παραθέσω κάτι από την εργασία του καθηγητή Γκούτχαρτ, που λέει ότι με κάποιους όρους που θα τους διαβάσω αν οι, αναπτυγμα... λέει, οι αναπτυγμένες κοινωνίες μπορεί να πρέπει να δεχθούν ότι η παραχώρηση κάποιας δημόσιας εγγύησης είναι ε, προϋπόθεση για λειτουργικό τραπεζικό τομέα. Και λέει, και άλλες μορφές ρυθμίσεων όπως διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις ε, και ε, με κυκλικότητα ε, αναλογία μόχλευσης ε, προς χρέωση για τη σταθεροποίηση των τραπεζών μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο με νέα ένταση. Οπότε ρωτώ τον κύριο Γκούντχαρ και τον κύριο Χέλβιτ, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ε, ότι τα, αυτά τα living wills και τέτοιες ρυθμίσεις είναι υποκατάστατα για τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις που ανέφερε ο κύριος Γκούντχαρ. Οι διαθήκες ζωής σε αυτά τα living wills έχουν δύο στοιχεία. Καταρχάς ε, την οδηγία για την ε, αναβάθμιση και ε, εξυγίανση των τραπεζών ε, και νομίζω ότι ένα καλό στοιχείο που είχαμε από την οδηγία αυτή είναι τα τεστ αντοχέ. Και τα τεστ αντοχή σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόγνωση. Αυτό που δείχνουν είναι ε, τράπεζες σε συγκεκριμένε συνθήκε που είναι πιο αδύναμες από άλλε. Και αυτό φυσικά μπορεί να αποτελέσει και το έναυσμα για να υποχρεωθεί μια τράπεζα να λάβει μέτρα ε, μάλλον αναβάθμισης πριν περάσει στην εξυγίαση. Και συνήθω τα θέματα τη εξυγίανση δεν ε, ξεκινούν παρά μόνο όταν η τράπεζα βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και όταν έχει ε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απολειών. Η, το πέρασμα από το bailout στο bail-in σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις απώλειες. Τι κάνει, συγκεντρώνει τις απώλειες απλώς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, μικρό αριθμό πιστωτών. Και αν αυτοί οι πιστωτές ε, είναι ε, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικέ εταιρείε, τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι συνέπειε για αυτού θα είναι ε, πάρα πολύ σοβαρέ και πολύ πολιτικά επιζήμιε, όπω και αν ήταν σε περισσότερου πιστωτέ. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τι ασφαλιστικέ εταιρείε από το να πρέπει να υποστούν αυτέ τι απώλειε, δηλαδή να κάνουν επενδύσει για διάσωση με ίδια μέσα, ε, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν, τότε κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ μικρός ε, ο πληθυσμός ε, του κυρίαρχου χρέους και των ταμείων που θα μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το χρέος. Σε καμία περίπτωση θα καταφέρετε μάλλον σίγουρα να πουλήσετε αυτά, αυτούς τους τίτλους ε, ε αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποτυχία, ιδίω όταν ε, ε, συμβεί όχι σε ιδιοσυγκρατικές συνθήκες, αλλά όταν υπάρχει περίπτωση μεγάλης πίεσης, τότε αυτό που θα γίνει είναι ότι θα... Ε, απομυζήσουμε κατευθείαν από την αγορά όλων αυτών των τίτλων ε, και αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλλες τράπεζες ή δεν θα είναι έτοιμες ε, να περάσουν και αυτοί τα κονδύλια που έχουν ε, αλλού ή θα έχουν έλλειμμα από το αποτελούμενο αποθεματικό. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πιέσεις για όλες τις άλλες τράπεζες και θα πρέπει οι άλλες τράπεζες να ε, δώσουν αποτελέσματα και σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιμόλυνση και ε, κυκλικά φαινόμενα από ό,τι έχουμε τώρα στο bailout. Και επομένως υπάρχει ένας δυνητικός κίνδυνος. Σε περίπτωση που έχουμε συστημική κρίση, η διαδικασία στην πραγματικότητα θα ενισχύσει την ε, επιμόλυνση και το συστημικό κίνδυνο και δεν θα τον προλάβει. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Συγγνώμη, ο κύριος Γκούτχαρτ στο έγγραφό του έλεγε ότι δεδομένων των παρατηρήσεων που κάνει, το θέμα της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης θα έρθει ε, στην πρώτη γραμμή και εδώ κάνουμε μία κρόση για την ε, ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Συγγνώμη, διακόπτει ο Πρόεδρος, είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα και δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι ομιλητές. Θα απαντήσουν στη συνέχεια. Το ECR. Ίσως θα μπορούσα ο κύριος Καμάλ να ε, συνεχίσω εγώ την ερώτησή σας. Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται τα τελευταία χρόνια είναι πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε σε λύσεις ώστε να αντλήσουμε διδάγματα και να μην έχουμε επανάληψη αυτών που έχουμε περάσει στο παρελθόν ε, στις πιο πρόσφατες τραπεζικές κρίσεις αλλά και στις προηγούμενες. Λοιπόν, έχουμε τρεις απλές προτάσεις τις οποίες εξετάζω. Πρώτον, πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να μην έχουμε ε, διάσωση με χρήματα των φορολογουμένων. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούν να αποτύχουν οι τράπεζες και δεν θα χρειάζεται να δώσουν χρήματα φορολογούμενοι. Αν όχι, ποιο είναι το όριο αυτής της παρέμβασης των φορολογουμένων και της ε, παρέμβασης με κεφάλαια. Όταν ε, χρεοκοπεί μια τράπεζα, κυρίως λιανικών ε, πωλήσεων, τότε θα υπάρχει πρόβλημα όταν κυρίως οι λιανικοί πελάτες δεν μπορούν μπορούν να πάρουν μετρητά από ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης ή από την τράπεζα. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει όταν μια τράπεζα κατά πάσα πιθανότητα ε, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, θα εξετάσουν καλύτερα τι γίνεται με το ισοζύγιο πληρωμών και να πούνε ότι αν αυτό ε, ε καταρρεύσει και εγώ είμαι υπεύθυνο, μήπως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλα όσα έχουμε στο ισοζύγιο πληρωνών μας. Και τέλος το θέμα των λογιστικών προτύπων. Οι τράπεζες μπορούν να έχουν ε, συγκεκριμένα προϊόντα στα ισοζύγια πληρωμών τους και από εκεί και πέρα μπορούν, θα πρέπει να δίνουν το εισόδημα ε, εκ των προτέρων χωρίς να προβλέπουν ε, επαρκώς τις απώλειες. Και στην πιο ακραία περίπτωση ε, αυτό που συνέβη με συγκεκριμένα δημοσιονομικά προϊόντα, ε, οικονομικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ε, ήταν ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Μήπως απομακρυνθήκαμε από τη σοφροσύνη και τα κατάλληλα λογιστικά πρότυπα και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητούμε σήμερα φαίνεται ότι από πολιτική σκοπιά φαίνεται ότι κάνουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν προσπαθούμε να λύσουμε τα πράγματα. Μήπως θα έπρεπε να σταθούμε σε πιο θεμελιώδη ερωτήματα, λογιστικά πρότυπα, ποιο έχει την ευθύνη ε, και το βασικό ερώτημα πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη διάσωση με χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Πώς αποφεύγουμε τη διάσωση, το bailout. Δεν τα αποφεύγουμε, είναι απάντηση η ανησυχία μου για την ε, οδηγία, για την εξυγίαση και την αναβάθμιση των τραπεζών είναι πολύ πιο θεμελιώδης ε, με του, από ότι του Φράνσις, του κ. Γκούτχαρτ, αλλά ε, με το Μπέιλιν διαφωνώ μαζί σου. μια τράπεζα σαν την BNP Paribas για παράδειγμα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες σε πάρα πολλές δικαιοδοσίες και η εξυγίανση θα σημαίνει ότι θα έχουμε πολλαπλές εισόδους και θα καταστρέψουμε την επιχειρησιακή ολοκλήρωση και κανένας δεν θα αναλάβει αυτό το κίνδυνο. Για εθνικά συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχει πρόβλημα ρευστοποίησης ε, στην εξυγίανση. Ε, η οδηγία δεν περιλαμβάνει τίποτα για το παροχή ρευστών και εδώ αναφερόμαστε σε 3 εκατομμύρια. Για πολλές τράπεζες μπορεί να είναι και 4 εκατομμύρια. Επομένως, στο βαθμό που αυτά είναι απλώς ανησυχίες, οι ε, κυβερνήσεις θα διασώσουν τις τράπεζες πολύ πριν φτάσουν στη διαδικασία της εξυγίανσης. Γι' αυτό και ίσως οι τίτλοι ε, τύπου Μπέιλιν μπορεί να μην μας ενδιαφέρουν καθόλου σε αυτή την περίπτωση ή μπορεί να αρνηθούν ότι υπάρχει πρόβλημα και να ελπίζουν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα επιλύσει το πρόβλημα στο μεταξύ. Και νομίζω λοιπόν εδώ ότι η διαδικασία που έχουμε, που είναι μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την απουσία διαδικασιών που είχαν κάποιες χώρες μέχρι τούδε, εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμη. Όσον αφορά την ευθύνη, νομίζω ότι ε, αυτό είναι ε, ε, κάτι το οποίο επιθυμούμε, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε και περισσότερες, περισσότερους τίτλους. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Τζάλ Σκούτχαρτ. Πολλά από τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή είχαν αντίστοιχα και πριν από το 2004 ε, διάφορες μορφές υβριδικών κεφαλαίων για παράδειγμα, τα οποία, οι οποίες ποτέ δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν και ο βασικός λόγος ήταν η πολιτική ισχύς και η πολιτική επιρροή των θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι επέβαλαν ουσιαστικά στις κυβερνήσεις τους να μην αφήσουν αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποτύχουν, να καταρρεύσουν. Και εδώ λοιπόν συμφωνώ με τις επιφυλάξεις του Τσάρλς, ε, ε, παρά το γεγονός ότι από πλευράς νομοθεσίας διαφωνώ μαζί του. Ευχαριστώ. Η Σιλβί Γκουλάρ τώρα. Συγγνώμη, δύο λόγια πρώτα. Ο κύριος Λίκα, ναι. Στην έκθεσή μας δεν υπήρχε το θέμα αυτό. Το βασικό ζήτημα που μας απασχόλησε και κυρίως ε, και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είχαμε φέτος στην Άνοιξη είναι ότι δεν έχουμε επιλύσει το too important to fail πρόβλημα και ε, στην πραγματικότητα οι εγγυήσει των κυβερνήσεων δημιουργούν κοινωνικές δυσκολίες διότι επιτρέπουν στις τράπεζες να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δημιουργούν περισσότερους κινδύνους. Ε, στην ομάδα εργασίας αυτή οι οποίοι μας έδισαν ε, ε, στοιχεία μας είπαν ότι ουσιαστικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να συνδυάσουν δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Από τη μια οι παραδοσιακές σχέσεις ε, ε, καταθέτει ε, και από την άλλη οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και θα μπορούσατε να ρωτήσετε ανθρώπους του κλάδου που θα σας πούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ Ισηβίγου Λάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να θέσω μια ερώτηση ε, που δεν είναι για πολιτικούς αλλά είναι πολιτικής φύσεως. Ποια είναι τα στρατηγικά σας ορέματα. Έστω ότι εγκρίνεται το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, ο κύριος Γκούτχαρτ λίγο πολύ μας απάντησε, και θα υπάρχει στρατηγικός έλεγχος στην Ευρώπη για αυτούς που χρηματοδοτούν την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί μόλις υπάρξει κρίση, εάν δεν έχουμε τρόπο να τα ελέγξουμε, οι αποφάσεις θα ληφθούν αλλού. Και το γεγονός ότι πρόκειται για μια στρατηγική παγκόσμια πρόκληση ε, μας δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα. Εγώ νόμιζα ότι ήμασταν κοινοβούλιο και ότι είχαμε εγκρίνει νομοθεσία, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι σε επιτροπές που δεν είναι μη ε, δημοκρατικές και μη νομιμοποιημένες, που έρχονται να μας πούνε αν είμαστε ε, συμμορφούμενοι με τον νόμο ή όχι και κάποιοι άλλοι που αναφέρονται ε, στο TILAC που προέκυψε εδώ και ξεπετάχτηκε σαν το μανεκτάρι. Ποια είναι η πολιτική στρατηγική σας και όχι η οικονομική. Ε, θα ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Ο κύριος Δεμάση τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους προσκεκλισμένους. Όταν, ήμουν, όταν σπουδάζα οικονομικά, έμαθα τον νόμο του Γκούντχαρτ και τώρα τον βλέπω μπροστά μου και μπορώ να του απευθύνω το λόγο απευθείας. Έλεγε ότι ό,τι κάνει στο χρηματοπιστωτικό τομέα ε, εφευρίσκεται μια καινοτομία για καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Πώς βλέπετε την σημασία της ρύθμισης τραπεζικού τομέα του σκιώδους και σε σχέση με τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στις τράπεζες. Βλέπετε να υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος ότι αν δεν είμαστε αρκετά αυστηροί με τις σκιώδεις κάποιες δραστηριότητες θα τις πάρουν αυτές. Δεύτερον, Ακούμε πολλά για την ε, Ένωση Κεφαλαιογοράσεων και ότι αν κάνετε τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και αν προχωρήσετε σε περαιτέρω ρυθμίσεις ε, ε, θα υπάρχει πρόβλημα με τη, τα, τη, τη δανειοδοσία. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Θέλετε πιο τραπεζοκεντρικό σύστημα ή υπάρχουν πλεονεκτήματα και από τη χρηματαγορά και κεφάλαια από εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα με την, τις πιστώσεις έχει να κάνει με το μακροοικονομικό περιβάλλον γιατί η ενδογενής ζήτηση ε, δανείων δεν είναι τόσο μεγάλη. Αναφέρεται τους ε, Lehman Brothers, τελειώνω, τελειώνω, που είχαν πρόβλημα. Οι Lehman Brothers δεν ήταν πρόβλημα διασύνδεσης μάλλον. Τι λέτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ποιος ήταν πρώτο, πρώτος ο κύριος Λίκανεν. Ε? Πολλοί μας ρωτούν για το όραμά μας. Το όραμα ήταν ότι οι τράπεζες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό ισχύει ακόμα. Είπαμε λοιπόν όλες οι τράπεζες καταθέσεων να έχουν το δικαίωμα όχι μόνο να δέχονται καταθέσεις αλλά να κάνουν και ε, αντασφαλιστικές διαδικασίες και να προχωρούν σε δανειοδοσίες. Ο μόνος τομέας, αν, αν κάναμε διαχωρισμό, θα ήταν αν προχωρούσαν πέρα από ένα ε, κατόφλιο. Οι τράπεζες λοιπόν θα παραμείνουν σημαντικές για την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, θα ήταν χρήσιμο για την ευρωπαϊκή οικονομία αν η, η, η, η θα αναπτυσσόταν περισσότερο γιατί έτσι θα υπήρχαν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης όπως γίνεται σε άλλες υπήρους. Και γι' αυτό στηρίζω την προσπάθεια στήριξης ε, της Ένωσης Κεφαλαίου Αγοράς ούτως ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Ο καθηγητής Γκούντχαρτ. Ένα πρόβλημα στην Ευρώπη ε, είναι ότι είναι υπερβολικά τραπεζοκεντρική. Ε, ε, δηλαδή ο χρηματοπιστωτικός τομέας περνά ως επιτοπλίστων από το τραπεζικό σύστημα. Θέλουμε κεφαλαία αγορά για διαφορετικότητα. Όσο μεγαλύτερη η διαφοροποίηση τόσο ασφαλέστερο είναι συνολικά το σύστημα. Ένα από τα προβλήματα με τις ρυθμίσεις είναι ότι είναι ε, εγγενώς προκυκλικές και ένας κίνδυνος είναι ότι ε, θα, αν γίνουν πολλά τα βήματα, τότε υπάρχει απομόχλευση και δεν αυξάνεται ο τομέας δανειοδοσίας. Και αυτό ε, δεν εξυπηρετεί την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, θα έλεγα η αγορά. Όμως ως ένα βαθμό οι ρυθμίσεις κεφαλαιακές που έχουμε, ιδιαίτερα το σύστημα στάθμισης κινδύνου, ε, είναι ε, ε, κατά αυτού του συστήματος. Τώρα θα πρέπει στις ισχυώδεις να έχουμε τα ειδικά hedge funds, ειδικά οχήματα και τα μία χρηματαγοράς. Τα ειδικά οχήματα και οι ρυθμιζόμενες τράπεζες έχουν να κάνουν με ρυθμιστικό αρμπιτράζ ή ε, τα ταμεία χρηματογοράς είναι το επικίνδυνο κομμάτι του συστήματος γιατί αυτές ε, ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με το... γιατί εκεί μπορεί να τρέξουν οι καταθέτες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Η Τραπεζική Ένωση, ε, τω μεταξύ, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού ε, ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αίσθηση των προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λάμπερτς. Καλό σας απόγευμα. Κύριε Γκούρθαντ, δεν είμαι βέβαιος ότι κατανόησα όταν είπατε πώς στοχεύετε να μας απαλλάξετε σε σχέση με τις εγγύσεις των φορολογουμένων ή μήπω το θεωρείτε αυτό σαν αγκαίο κακό. Θα ήθελα να το κατανοήσω καλύτερα, να το διευκρινίσετε και συνδέεται με αυτό. Αν αυτό είναι αναγκαίο κακό, ήθιστε να συμβαίνει σε μια οικονομία της αγοράς οι προοπτικές που συνδέονται με τις επιδοτήσεις να ιδιωτικοποιούνται και οι παρέχοντες αυτές τις εγγυήσεις, δηλαδή οι φορολογούμενοι, τα συστήματα αυτά θα εθνικοποιούνται σε σχέση με τα κόστη και τα κέρδη για την παροχή των επιδοτήσεων και σε όλους σας ερώτημα για την τράπεζα φόρτης ε, της, ε, του Βελγίου. 45 δις τοξικά προϊόντα είχε αυτή η τράπεζα και υποχρεώθηκε να, ε, αν υποχρεωνόταν να διατηρήσει τις διαστηριότητες της ε, ξεχωριστά, θα γινόταν μια ξεχωριστή τράπεζα και δεν θα μπορούσε να έχει τα 45 δίσα ε, σε τοξικά προϊόντα πλέον. Δηλαδή όλα αυτά το, ε, σε σχέση με αυτά τα προϊόντα με βάση την ζήτηση, ίσως σε σχέση ακριβώς με την προσφορά και τη ζήτηση να μπορείτε να διευκρινίσετε κάτι. Ευχαριστώ. Μάρκο Τζάνι, επόμενο αγορητή, παρακαλώ. Ναι, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του ομιλητέ μας. Εγώ νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε διαρθρωτική μεταρρύθμιση ε, του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να θέσουμε δύο βασικές ερωτήσεις για να κατανοήσουμε τι λύσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε, να περιορίσουμε τον ηθικό κίνδυνο από πλευράς τραπεζών που κατά πάσα πιθανότητα ήταν το πρώτο αίτιο των τραπεζικών κρίσεων που βιώσαμε και κυρίως ε, την κρίση του 2008. Δηλαδή την ακραία αναζήτηση μεγιστοποίησης του κέρδους ε, μέσω οποιοδήποτε προϊόντος. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες θα ε, αρχίσουν και πάλι να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Επομένως θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δομή κατά την άποψή σας που είναι η ιδεώδης προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο και αν θεωρείτε πραγματικά το, ότι το μοντέλο της ε, τράπεζας ε, γενικών διαδικασιών είναι πραγματικά το ιδανικό μοντέλο για να επιτευχθεί αυτό ο στόχος. Αν είμαστε πεπισμένοι ότι μόνο μέσω διαχωρισμού και διάσπασης των τραπεζιών μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό, ε, δεδομένου ότι και διαρθρωτικά εδώ και κάποια χρόνια οι τράπεζες ήδη εγκαταλείπουν κάποιες δραστηριότητες ε, χρηματιστηριακές. Ε, μια ακόμα γρήγορη ερώτηση για τα παράγωγα, δεδομένου ότι αποτελούν πολύ μεγάλο κίνδυνο ούτω ή άλλως ε, για τους ισολογισμού των τραπεζών. Μήπως θα έπρεπε στη μεταρρύθμιση αυτή να καθορίσουμε και κάποια ανεξάρτητη αρχή, όπως ε, η αρχή που συστάθηκε στις ΗΠΑ ε, το 2008, που να προσπαθήσει να αξιολογήσει του κινδύνου των ε, με βάση τι μεγαλύτερε Ευρωπαϊκέ Τράπεζε. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση απευθύνθηκε προς τον καθηγητή Γκούτχαρ. Ε, Επομένω θα ξεκινήσουμε από εσά. η επιδότηση ε, σε γενικές ε, τράπεζες που είναι σημαντικές συστημικά θα είναι κάτι αναπόφευκτο και μάλιστα περισσότερο σε αυτές τις τράπεζες από ό,τι άλλες και υπάρχουν τράπεζες νομίζω οι οποίες θα προτιμούσαν να μην υπερβαίνουν αυτό το κατώτατο όριο και να θεωρηθούν ότι είναι σημαντικές ε, ε, συνολικά. Θεωρώ ότι είναι λογικό οι μεγαλύτερες τράπεζες που θα ε, δημιουργήσουν μεγαλύτερες ζημίες όταν καταρρεύσουν θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες κεφαλαιακές αποτίσεις και αυτό φυσικά σχετίζεται και με το θέμα της ενίσχυσης. Όσον αφορά τον ηθικό κίνδυνο, ε, πρόκειται για μια φράση που ε, χρησιμοποιείται παραπάνω συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Οτιδήποτε προστατεύει τους ανθρώπους ενάντια σε ε, επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνει κάποιο ηθικό κίνδυνο. Επομένω, οτιδήποτε προσπαθεί να κάνει ασφαλέστερο το, το σύστημα ενέχει κάποιο ηθικό κίνδυνο. Και νομίζω ότι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις έχουν κίνητρα τα οποία θα έχουν σταθμίσει δεόντως. Δηλαδή να δουν την ε, δομή ε, μισθοδοσίας των ε, υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών. Ευχαριστώ. Εσείς ένα σχόλιο έχω μόνο για το πώς οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η διάθεση δηλαδή δανείων θα μπορεί να είναι κερδοφόρο δραστηριότητα και γι' αυτό το κάνουν οι τράπεζες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό γίνεται με φθηνό τρόπο, χωρίς κόστη. Και υπάρχουν λοιπόν πολιτικές επιέσεις για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν θέλετε να επιδοτήσετε όμως, καλύτερα θα ήταν να επιδοτούνται άμεσα διαφορετικά να τα αφήσει κανείς σε κερδοφόρες δραστηριότητε τραπεζικές, χωρίς όμως να εισάγονται στρεβλώσεις σε σχέση με τους ισολογισμούς των τραπεζών με βάση τις διατάξεις για την διάθεση κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Λίκανε. Για την ερώτηση για τη φόρτιση δεν απαντήσατε όμως. Για το θέμα για συγκεκριμένες τράπεζες αν είχα χρόνο θα μπορούσα φυσικά να το κάνω αυτό, αλλά είναι ταχύτατη η ανάπτυξη αυτών των τραπεζών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και στις ε, συναλλαγές ε, ή στην υπερβολική δανειοδότηση. Η υπερβολική δανειοδότηση, συμφωνώ με τους συναδέλφους, ήταν ένας κίνδυνος. Τώρα, με τον κύριο ε, Γκούτχαρντ, συμφωνώ ότι είναι κέρια σημασία αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι αν υπάρχει στην ίδια τράπεζα διτή δραστηριότητα, συναλλαγές γενικού ε, κερδοφόρου χαρακτήρα, που μακροπρόθεσμα σε σχέση με δανειοδότηση δεν ε, έχουν τα ίδια κέρδη. Ε, και παραδοσιακά μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν και πολλές μεγάλες τράπεζες ε, που έδωσαν ε, τα στοιχεία ότι σε σχέση με την, τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων εγώ πιστεύω ότι η σωστή χρηστή διακυβέρνηση είναι εκείνο το οποίο μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για τη διαδικασία Καστιάη με αγορίτες. Ίσως στο τέλος θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε αν υπάρχει χρόνος Τώρα πρέπει να δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Yes. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο χρόνος πιέζει και καλό θα ήταν να είχαμε τη διαδικασία Κατσδιάη. Ένα πράγμα όσον αφορά τις ε, επιδοτήσεις. Πιστεύω ότι με οποιοδήποτε τρόπο και αν αξιολογήσουμε αυτό, τουλάχιστον ε, η εμβέλεια αυτού του ε, φαινομένου ε, έχει, μπορεί να μειωθεί. Τουλάχιστον όταν υπάρχει το φαινόμενο αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και ένα άλλο πράγμα, μια άλλη πτυχή. Και έχει γίνει αναφορά σε αυτό οι επενδυτικές τράπεζες ή οι τράπεζες γενικών ε, εργασιών έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια δραστηριοτήτων, πολυσχυδέστερες δράσεις από ότι οι τράπεζες καταθέσεων. Και πιστεύω ότι για να καταφέρει κανείς να διασφαλίσει την αξιοπιστία όσον αφορά τέτοιου είδους συναλλαγές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να πει κανείς ότι οι ε, τράπεζες ε, αυτών των ε, λιανικών εργασιών είναι ασφαλέστερες όταν έχουμε το θέμα του bail-in. Γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ πιο περίπλοκο πλέγμα στην ίδια την πραγματικότητα όταν έχουμε το θέμα bail-in από πλευράς κεφαλαίων. Αυτό προτού δοθεί οποιαδήποτε συνέχεια σε αυτό. Ευχαριστώ. As Δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσει ο πρόεδρος και εγώ θα προεδρεύσω μέχρι τέλους. Ξεκινάμε το δεύτερο πάνελ αγόριτων για τις επιλογές διαφορετικών δυνατοτήτων μεταρρυθμίσεων. Υπενθυμίζω ότι 7-8 λεπτά θα είναι ο χρόνος ε, και παρακαλώ να μην έχετε ταχύ ρυθμό εκφοράς ε, γιατί προβλέπεται να ολοκληρωθεί αυτό το πάνελ στις 6 ε, και 25 ή προς 6 και 30. Ξεκινάμε αμέσως λοιπόν με το πάνελ αυτό. Πρώτος αγορητής, ο καθηγητής Μάρκο Παγκάνο πρόεδρος ε, της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και επίσης έχει ε, συμβουλέψει την ΕΣΜΑ και το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσίασή μου σύντομα θα προσπαθήσει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των ε, ε, δομών των ε, τραπεζών. Ποιες μεταρρυθμίσεις μπορούν να, αναμένονται και με ποια ωφέλη. Πώς θα, θα επιμεριστεί το κοινωνικό κόστος όσον αφορά την, τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Για τα κοινωνικά ωφέλη που μπορούμε να αναμείνουμε με την επιβολή περιορισμών όσον αφορά τη δομή τραπεζών, όπως ήδη ακούσαμε από τους προλαλήσαντες αγορητές. Το πρώτο όφελος είναι η μείωση συστημικών κινδύνων που επομίζονται οι τράπεζες και το δεύτερο μείωση των, ε, ε, των ε, εγκυοδοτήσεων όσον αφορά την ρίση του big to fail. Γιατί μπορούμε να αναμένουμε αυτά τα ωφέλη. Για δύο λόγους. Απουσία των μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει στο να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στις δανειοδοτικές δραστηριότητες σε εταιρείε, σε νοικοκυριά και σε άλλους. Εξού λοιπόν έχουμε μια ευρεία βάση και ε, μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων ε, στην οικονομική δραστηριότητα αφενός και στην σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. Έκθεση δηλαδή σε ε, μολυσματικούς κινδύνους. Κάτι τέτοιο ως μεταρρύθμιση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης και μπορεί να αυξήσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ένας άλλος λόγος που μπορούμε γι' αυτό να αναμένουμε ωφέλη είναι ότι θα μπορούν τα επιτόκια να, απο, να δημοσιοποιούν το τι συμβαίνει σε σχέση με τις ε, επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις και μειώνοντας ε, ή περιορίζοντα περιορίζοντας ε, τις α, επιδοτήσεις αυτές και ιδιαίτερα όσον αφορά τις Αυτά, αυτού του είδους τα ωφέλη θα είναι ε, ιδιαίτερης εμβέλειας και θα πρέπει να στοχεύουν και τις μεγαλύτερες τράπεζες, διότι αυτές οι τράπεζες εκτίθενται περισσότερο και δραστηριοποιούνται στις επενδυτικές δραστηριότητες και εκτίθενται σε σχέση με τους, ε, όσους διαμεσολαβούν σε αυτές τις συναλλαγές και μια κατάρρευσή τους θα είχε ε, αρνητικότατες επιπτώσεις. Και αυτό βλέπουμε σε σχέση με την έκθεση ε, του 2014 που δείχνει ότι οι συστημικοί ε, κίνδυνοι συνδέονται με το μέγεθος ε, και με το είδος το, το είδος δραστηριοτήτων που ακολουθεί μια τράπεζα. Και έτσι λοιπόν με, τον, με την μείωση των συστημικών κινδύνων από τις μεγαλύτερες τράπεζες θα είναι εκείνο το οποίο θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε και σε σχέση με όσους εκτίθενται περισσότερο σε εμπορικές συναλλαγές και όχι τόσο σε δανειοδοτήσεις. Τώρα, σε σχέση με το σχεδιασμό της μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα, το να πετύχουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις ε, ώστε να ε, ξεχωριστούν ε, οι δραστηριότητες οι τραπεζικές από, τους, από τις συναλλαγές που συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους. Αν πάρουμε το σχέδιο οδηγίας, δηλαδή τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων σε δύο ε, μονάδες, ε, σε ε, μία μονάδα συναλλαγών και μία άλλη μονάδα ασφαλέστερων δραστηριοτήτων, μπορούμε να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης εξαρτάται από τρία σημεία που αφορούν την ποιότητα των συναλλαγών για την δυνατότητα ορίων που πρέπει να επιλεγούν για την, ε, τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων. Δεύτερον, ποιες εξαιρέσεις ε, θα ε, ισχύουν για κάποιες δραστηριότητες δανειοδότησης, παράδειγμα κρατικό χρέος και δεύτερον, Ποιο θα είναι το επιτρεπόμενο μέγεθος για τις, την έκθεση τέτοιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών βλέπουμε ότι οι κυριότερες δραστηριότητες που μπορούν να, διαχωρίζονται από τις ε, ε, πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες, αν δεν υπάρξει ε, σαφής διαχωρισμός, τότε θα είναι λιγότερο επιτυχής η μεταρρύθμιση. Και γι' αυτό ας ε, επανέλθω στο θέμα το οποίο βρίσκεται στην ίδια τη συζήτηση ως βάση. Ανάπτυξη. Όταν εξετάζουμε τη μεταρρύθμιση πρέπει να δούμε ε, αν αυτό θα μείωνε την δανειοδότηση σε σχέση με επιχειρήσεις και νοικοκυριά ενώ ίσως ε, αυτό θα μπορούσε να αναφέρεται στην σημερινή συγκυρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η ανησυχία νομίζω δεν, δεν ευσταθεί αυτό το οποίο συμβαίνει σε σχέση με το 2014 στην έκθεση που αναφέρεται, ο τραπεζικός τομέας ε, έχει φτάσει ε, σε ένα μέγεθος που δεν συνεισφέρει πλέον θετικά στην οικονομική ανάπτυξη. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι πέρα από ένα κατόφλι του ΑΕΠ, μια, ένας, μια θετική αντιστοιχία, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο, ε, πάβει να υπάρχει και μάλιστα ακολουθεί μια ευθύνουσα τάση. Και θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να ε, κατευθυνθούμε προς ε, τον τομέα των ε, ακινήτων και την χαμηλότερη παραγωγικότητα και τη μεγαλύτερη εμβέλεια σε λιγότερο παραγωγικές δραστηριότητες. Η ε, έκθεση η τραπεζική της ε, SRB δείχνει ότι οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν από τις μεγαλύτερες τράπεζες, διότι αυτές θα υφίστανται τις επιπτώσεις ε, του διαχωρισμού αυτού. Πράγματι, αν οι μεγαλύτερες 20 τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε σχέση με το 1996 αντιστοιχιστούν, το 2012 θα είχαμε περίπου το ίδιο ποσοστό ΑΕΠ όπως το 1996 ο διπλασιασμός σχεδόν μπορεί να πούμε ότι αντισταθμίζεται από την ανάπτυξη των μεγαλύτερων τραπεζών. Και για την ρευστότητα των αγορών, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ο φόβος ότι το πιθανό κόστος αυτής της μεταρρύθμισης θα οδηγήσει στο ότι οι μεγαλύτερες ε, ε, τράπεζες ε, να πρέπει να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ωστόσο όμως αυτό νομίζω υπερβάλλει για τους εξής λόγους. Πρώτον, η πρόταση για, την, για του είδους αυτό ε, των συναλλαγών υποτιμά τις δυνατότητες. Δεύτερον, η μείωση των ε, αγορών ε, ασφαλίσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί με την παροχή ρευστότητας από άλλες δραστηριότητες σε σχέση με την δυνατότητα να μπορεί να επιδοτείται η δραστηριότητά τους με την αρχή too big to fail και την εγγύηση που αυτό θα συνεπαγόταν. Ε, οι άλλες ε, ε, δυνατότητες για διαμεσολαβητές σε σχέση με κατακαιρματισμένες αγορές που οδηγούν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο κεντρική κεντρι κεντρικής δομής αγορές με ηλεκτρονική λειτουργία. Και αν εδώ υπάρχει το θέμα της ε, επιδότησης, υπάρχουν πολύ πιο άμεση τρόποι και πιο διαφανείς τρόποι να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ε, έμεσα με τις ε, διασταυρούμενες επιδόσεις από τις μεγάλες τράπεζες υπό την αρχή του big to fail. Αυτές ε, οι έμεσες επιδοτήσεις ε, συνεπάγονται όμως κοινωνικά επιβλαβείς ε, επιπτώσεις καθώς επίσης και τις, τα φορολογικά θέματα τα οποία όλα αυτά θα συνεπαγόντουσαν. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, ευχαριστώ καθηγητή Παγκάνο. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο μιλητή μας. Η κυρία Πρεσβόσκα που είναι αναλύτρια στο Finance Watch. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, σας δίνω το λόγο. Είναι τιμή για μένα να βρίσκουμε εδώ ως αναλύτρια του Finance Watch και να σας παρουσιάσω την έκθεσή μας. Ε, λόγω των πιέσεων ε, των χρονικών θα ήθελα να σταθώ στις συνέπειες μιας αποτελεσματικής διαρθρωτικής μεταρρύθμισης από χρηματοπιστωτική πλευρά. Αν είχα τρία πράγματα μόνο να σας πω θα ήταν το εξής. Πρώτον, αποτελεσματική μεταρρύθμιση των τραπεζών σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους συστημικού κινδύνους, έχει μακροοικονομική εστίαση και ενδιαφέρεται για συγκεκριμένα ε, καθεστώτα όπως κεφαλαιακές απαιτήσει και εξυγίαση. Αυτό λαμβάνουν υπόψη ε, ε, βέβαια ε, μόνο κάποιες αδυναμίες και δεν ε, καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν συστημικούς κινδύνους. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος επιμόλυνσης από τις ε, εμπορικές δραστηριότητες, τις βασικές δραστηριότητες των συστών. Αυτές λοιπόν οι βασικές δραστηριότητες πρέπει να προστατεύονται και πρέπει να καλύπτονται από ένα βασικό δίκτυο ασφαλείας. Και τέλος, η μετα... μεταρρύθμιση θα πρέπει να εστιάσει στις αδυναμίες του τραπεζικού μοντέλου δεν θα πρέπει να απειλεί τις μικρομεσαίες ε, ε, τράπεζες γενικών εργασιών. Το αντίθετο θα πρέπει να ενισχύσει την ε, πειθαρχία της αγοράς. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με το παράδοξο τώρα των ρυθμιστών για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ε, υπάρχει ε, ένα κοινό κεφάλαιο το οποίο χρειαζόμαστε ακόμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την πραγματική οικονομία. Όμως οι ε, τράπεζες ε, αυτές οι οποίες είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν χρειάζονται πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό ε, δεν επαρκεί για να μπορέσει να τους προστατεύσει και σε ...περιγράφηκε σε κάποια εργασία ε, του αντρερ Μπλούντεν Βίγκελ και του Πολ Άτκισον και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη διαστατική μεταρρύθμιση. Ε, η άποψη της Finance Ones είναι ότι μια αποτελεσματική διαστατική μεταρρύθμιση θα πρέπει να προστατεύει από τις, τις βασικές ε, τραπεζικές δραστηριότητες από εξε, υπερβολικούς κινδύνους και υπερβολική εμπορία και κυρίως εμπορία παραγόγων. Μπορεί να φέρετε πλέον κάτι πολύ απομακρυσμένο. Το 2008 πραγματικά υπήρχε φόβος κατάρρευση της κοινωνίας. Και γιατί αυτό, διότι ε, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των στρατηγικών, γιατί και οι δύο στρατηγικές απαιτούν ε, να υπάρχουν κεφάλαια για να προστατεύσουμε τις βασικές ε, δραστηριότητες. Ε, οι βασικές δραστηριότητες θα πρέπει να μένουν ίσως στις ίδιες ομίλου τραπεζών ε, για λόγους συνέργειας, αλλά δεν θα πρέπει οι πιστωτές ε, του πιστωτικού ιδρύματος να μπορούν να πάρουν στοιχεία ενεργητικού για να τα χρησιμοποιήσουν για εμπορία παραγόγων. Ε, και αυτά φυσικά θα πρέπει να τα προστατεύσουμε στην ενιαία αγορά. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες τώρα για τις συνέπειες μιας αποτελεσματικής διευθυντικής μεταρρύθμισης και κυρίως θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στις συνέπειες για το κάθε τραπεζικό ε, ίδρυμα και θα πρέπει να λάβουν υπόψη και το ιδιωτικό κόστος. Οι συνολικές συνέπειες δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη. Εδώ τώρα θα ήθελα να σταθώ λίγο στις ε, ε, διαβόητες αρνητικές συνέπειες μιας αποτελεσματικής μεταρρύθμισης. Οι πρώτες ανησυχίες είναι ότι το σύστημα ε, των γενικών τραπεζών θα ζημιωθεί αν γίνει μεταρρύθμιση, ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση ε, και η διαφοροποίηση για το πλεονέκτημα θα ε, χαθεί και θα χαθούν και οι οικονομίες κλίμακας. Το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης είναι μεγάλο και κατάλληλα συγκεντρωμένο σε πολύ συγκεκριμένα. Αν δούμε συγκεκριμένα στοιχεία ρεστοποίησης τράπεζας, θα δούμε ότι υπάρχουν συγκέντρωση γύρω από 20 μεγαλύτερες τράπεζες και από τον υπόλοιπο τομέα. Υπάρχει λοιπόν σαφής διάκριση μεταξύ αυτών και υπάρχει λοιπόν αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο για τις τράπεζες που είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν, αλλά δεν επιδρά αρνητικά στις μικρές και μεσαίου μεγέθους τράπεζες γενικών εργασιών. Και ε, το θέμα είναι ε, ότι μέχρι την κρίση οι τράπεζες που είχαν διαφορετικές ε, επιχειρηματικές γραμμές υποτίθεται ότι θα αποφελούνταν από τη διαφοροποίηση αυτή. Αλλά ένα χρηματοοικονομικό σύστημα στο οποίο η κάθε τράπεζα φαίνεται ότι είναι υγιής μπορεί να είναι ασταθές όταν εκτίθενται σε κοινού κινδύνους. Και οι ψηλά διαφοροποιημένες γενικές τράπεζες μπορεί να σχετίζονται η μία με την άλλη και να δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο μιας κοινή τραπεζικής κατάρρευσης. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα υγιές ε, μακροοικονομικό ε, σύστημα το οποίο θα είναι και κατάλληλα προληπτικό για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αλλά και να ελέγξουμε αυτούς τους κινδύνους θα υπάρχουν μόνο συγκεκριμένε επιδοτήσεις ε, ε, για, τις, ε, για την εμπορία που θα εξαφανιστούν, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε και τα θετικά αποτελέσματα αυξανόμενου ανταγωνισμού και περιθασμίας της αγοράς. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που καταδεικνύουν ότι όταν λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες ενισχύσεις, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι οικονομίες κλίναβας εξαφανίζονται. Δεύτερον, λέγεται ότι δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμες οι εμπορικέ δραστηριότητες και οι υπηρεσίες θα είναι πολύ πιο δαπανηρές για πελάτες και ε, μπορεί εμπορικέ δραστηριότητες να εξαφανιστούν από την αγορά. Εγώ συνήθως απαντώ ε, με το πώς ε, το σύστημα το επενδυτικό των τραπεζών άνθησε με βάση τον νόμο Glass-Steagall. Και πραγματικά δεν θα χρηματοδοτείται ο εμπορικός κλάδος από ε, τον αποτελεσματικό διαχωρισμό και σημαίνει ότι αυτές οι δραστηριότητες θα είναι κατάλληλα διαχωρισμένες και θα μπορεί να υπάρχει κατάλληλη ε, τιμολόγηση που θα μας βοηθήσει να έχουμε ε, οικονομική σταθερότητα. Ολοκληρώνοντας, το γεγονός ότι συζητάμε πώς θα εφαρμόσουμε τη στρατιωτική μεταρρύθμιση και όχι κατά πόσον θα την, πρέπει να την εφαρμόσουμε, καταδεικνύει ότι τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη μεταρρύθμισης και αυτό είναι θετικό, αλλά θα πρέπει να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική για να μπορέσει να δημιουργήσει τι αλλαγέ που χρειάζονται. Εάν ε, τα κατώτατα όρια είναι πάρα πολύ γενναιόδερα και ε, ο φράχτη είναι πάρα πολύ χαμηλό και υπάρχει πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια, η διαστατική μεταρρύθμιση των τραπεζών ελοχεύει ο κίνδυνο να γίνει απλώ ένα γραφειοκρατικό μέτρο. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο Καντέρα από την BBBA. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γιατί απεδέχθη μια καθυστερημένη πρόσκληση ε, για να αντικαταστήσει έναν ομιλητή που δεν μπόρεσε να μείνει. Εργάζεται για μια μεγάλη ε, τράπεζα γενικών εργασιών. Κύριε Κρέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτό το θέμα. Όχι μόνο εξ ονόματος του δικού μου Ιδρύματος, Μεγάλη Ισπανική Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και εξ ονόματος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ε, για ε, τις τραπεζικές εργασίες. Σκοπό έχω να εξηγήσω γιατί η πρόταση της Κομισιόν για την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των ε, τραπεζών δεν χρειάζεται, δεν δικαιολογείται. Θα μιλήσω για τρία βασικά θέματα. Ε, το θεματολόγιο της ε, ρύθμισης, το ρόλο των γενικών τραπεζών και τον αντίκτυπο του προτινομένου κειμένου. Καταρχήν θέλω να σας μιλήσω για τα ευραία μέτρα που έχουν ληφθεί, που συζητούνται από τους ρυθμιστικούς φορείς ευρωπαϊκούς και ε, παγκόσμιους. Πάνω από 40 πρωτοβουλίες μεταρρυθμιστικές έχουν εγκριθεί από το 2008 ήδη πιο κυρίες είναι η μόχλευση, το ιδέσμι για τη ρευστότητα, τα κεφάλαια και η οδηγία για την εξυγένση των τραπεζών που δίνει τη δυνατότητα στους ρυθμιστικούς φορείς να αλλάξουν τη διάρθρωση της τράπεζας για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και φερεγγιότητα. Ε, επίσης ελήφθησαν πρωτοβουλίες και σε παγκόσμιο επίπεδο για να ενισχύσουν την αγορά παραγόγων και να ε, ε, ε, αναθεωρήσουν την διαδικασία διαπραγματεύσεων. Σημαντικό είναι οι συστημικές τράπεζες να αντέξουν την κρίση. Αυτές αντιμετωπίζονται με το «do big to fail. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ε, και ο νέος επόπτης για την Ευρωζώνη ε, σηματοδοτεί μια μετατόπιση στην εποπτεία τραπεζών. Η εποπτεία τώρα γίνεται πιο συγκεντρωτική, πιο εντατική, πιο αποτελεσματική και πιο αποφασισμένη ε, για να αναλάβει αποφασιστική δράση. Τώρα, δύο λόγια για τις τράπεζες γενικών εργασιών. Η Γενική Τραπεζική είναι ένα πλεονέκτημα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος και η έρευνα που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι η διαφοροποίηση εσόδων που προέρχεται από αυτήν ε, κάνει τις γενικές τράπεζες να είναι σε καλύτερη θέση για να στηρίξουν τους πελάτες τους ε, τους, ε, της ΜΜΕ σε περιόδους οικονομικής κάμψης είναι κλειδί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δηλαδή. Το μοντέλο της Τράπεζας Γενικών Εργασιών ε, φάνηκε να είναι από τα πιο ανθεκτικά ε, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γεγονός ότι πολλές μικρότερες τράπεζες διασώθηκαν κατά την κρίση δείχνουν ότι τα, οι περιορισμοί στο μέγεθος δεν αποτελούν πανάκια. Πρέπει να θυμηθούμε ότι οι γενικές τράπεζες δεν παρέχουν μόνο υπηρεσίες ε, στο λιανικό εμπόριο και στις ΜΜΕ, αλλά είναι πηγές ρευστότητας και συνδεδεμένων υπηρεσιών για τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης, όπως είπε η έκθεση στην γνωμοδότησή της για την ε, πρόταση της Κομισιόν, είναι θεμελιώδες να διατηρηθούν οι δραστηριότητες στην αγορά για να διατηρούνται ή να αυξάνονται τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, η ρευστότητα, ε, οι διακυμάνσεις και να υπάρχει ε, αντοχή της αγοράς στα σοκ. Η έκτη υπογραμμίζει επίσης ότι ε, είναι σημαντική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα η ε, λειτουργία της αγοράς ε, για την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής και τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Όπως όμως αναφέρεται, η αρχική πρόταση θα επηρεάσει αρνητικά το κίνητρο των γενικών τραπεζών να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες market making. Έτσι, οι ρευστότητες της αγοράς ε, θα μειωθεί σε ορισμένα μέσα ε, και έτσι η χρηματοδότηση θα δυσχερανθεί. Ε, θα μειωθεί, αν μειωθεί ο ρόλος των τραπεζών θα υπονομευθεί η Ένωση Κεφαλαίου Αγοράς ως εναλλακτική για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Η αρχική πρόταση για τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών είναι... θα πρέπει να συζητηθεί με τους εμπλεκομένους. Πριν προχωρήσω σε συμπεράσματα, θέλω να υπογραμμίσω κάποιες επιπτώσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά τις διαχωρισμένες μονάδες ε, στις διαπραγματεύσεις, στις συναλλαγές ε, θα είναι μεγαλύτερο το χρηματοδοτικό κόστος. Υπολογίζεται η αύξηση του κόστους ε, στο, στα 220, 220 μονάδες 2,2%. Μια τέτοια αύξηση θα μειώσει τη δυνατότητα ε, παροχής υπηρεσιών αγοράς. Όπως αναφέρεται στην νομοδότηση της ΕΚΤ, διαχωρισμός από μόνος του δεν λύνει το θέμα του big to fail και οι συνέπειες του υποχρεωτικού διαχωρισμού θα είναι συγκέντρωση υπηρεσιών προς τους πελάτες σε, στα χέρια λίγων παικτών στην αγορά. Ο αυξημένος ανταγωνισμός από μη ενωσιακό ιδρύματα και η μείωση της ρευστότητας στις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ε, προαπαιτούμενα στους, ε, των πελατών ΜΜΕ, δηλαδή ε, συναλλαγές ειδικέ, το Ίδρυμα που στηρίζεται σε κρατήρια επιχείρησης θα ε, ε, ε, μειώσει τη δυνατότητά του να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Αυτό με τη σειρά του θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά των ΜΜΕ. Επίσης, το κόστος χρηματοδότησης για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα επιδράσει αρνητικά στη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να επανεξεταστεί η τωρινή πρόταση. Η επανεξέταση πρέπει να λάβει υπόψη τον έντονο μετασχηματισμό ε, των τραπεζικών πλαισίων ε, ε, εποπτείας και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Κομισιόν για διατηρήσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας μας και περαιτέρω ανάπτυξη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κεφαλαία αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εσάς κύριε Κρέμα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Και το βλέπει κανείς και από τα πρόσωπα των ε, όσων σας παρακολουθούσαν. Και τελευταίος αγορητής, ε, ο κύριος Dirk Βάουτερς, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, των Τραπεζών, για να μας δώσει την δική του παρέμβαση για αυτό το θέμα. Κύριε Βάουτερς, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας για την ευκαιρία που παρέχετε και με αυτή την πρόσκληση να έρθουμε ενώπιον σας. Ε, το εκτιμούμε ότι οι μικρές τράπεζες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση για το, τις δραστηριότητες. Ε, ποιες εμπορικές δραστηριότητες ε, είναι ουσιώδους χαρακτήρα για τις τράπεζες ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Μικρές τράπεζες που εξειδικεύονται στις ε, διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες ε, έχουμε εξειδικευτεί στην χρηματοοικονομική διαφορά μέσω των ε, δραστηριοτήτων μας που εξακολουθούν και υφίστανται, που, μπορεί όμως παρόλα αυτά να είναι περιορισμένες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βοηθούμε τους πελάτες μας. Ε, ένα μικρομεσαίο για παράδειγμα που ε, έχει κάποια πληρωμή ε, που θα γίνει μετά από 6 μήνες και θέλει τα επιτόκια να καθοριστούν αυτή τη στιγμή. Καθορίζουμε και βοηθούμε λοιπόν για τον υπολογισμό των επιτοκίων και πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά τα κονδύλια με τους ομολόγους μας. Όμως δραστηριοποιούμαστε ένεργα βοηθώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το επιχείρημα το ότι οι διαφορετικές ε, αλλαγές ε, θα παρακολύσει τις τράπεζες ε, να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στους πελάτες τους δεν με πείθει. Έχουμε μικρότερη εμβέλεια σε σύνθεση όσον αφορά τους πελάτες μας όταν έχουν καθοριστεί τα προαπαιτούμενα πάμε στις χρηματοοικονομικές αγορές για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Αυτό συνεπάγεται φυσικά ότι από πλευρά μα ε, οι αμοιβέ ε, σε σχέση με τον ε, κειμενόμενο χαρακτήρα που μπορεί να έχουν πρέπει να διασφαλίζονται αποκλειστικά από τις δραστηριότητες μας αυτές, αυτών των συναλλαγών. Αν θέλουμε να προστατέψουμε αυτή τη θέση μας μέσω συναλλαγών πελατών μας χρειαζόμαστε μια ρευστή αγορά. Χρειαζόμαστε άλλους εμπλεκόμενους στην αγορά, μεγαλύτερες εμβέλειας για την παροχή ρευστότητας που είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν το παιχνίδι στην αγορά. Ενώ είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίζει κανείς ε, τη δημιουργία τέτοιων ευκαιριών ε, σε σχέση με την ε, δυνατότητα παροχής ρευστότητας, νομίζω μπορεί να επιτευχθεί αυτό Δηλαδή σε σχέση με την πρόταση να δώσουμε στην ε, εξουσία της εποπτικές αρχές ε, να καθορίσουν κάποια όρια θα ήταν μια καλή ιδέα και ας μην ξεχνάμε ότι οι δραστηριότητες ε, της παροχής ρευστού έχει τις ρίζες της στην ίδια τη ζήτηση από την αγορά και την ζήτηση από πελάτες που θέλουν να εξασφαλίσουν τις ε, δραστηριότητες τους ε, με τις θέσεις ε, που έχουν τραπεζικά. Και μέσω των εμπορικών αυτών δραστηριοτήτων και συναλλαγών και για την διασφάλιση ρευστών δεν ε, είναι ε, η δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών τόσο όσο η ζήτηση ρευστότητας που υφίσταται και νομίζω μπορεί να διοργανωθεί σε συνετά πλαίσια αυτό. Όσον αφορά τώρα την διαχείριση κεφαλαίων, οποιαδήποτε τράπεζα δραστηριοποιείται σε εμπορικές συναλλαγές κύριος ε, πυρήνας ε, των ε, εργασιών των τραπεζών είναι οι καταθέσεις τα διαθέσιμα αποθεματικά να μπορούν να διατεθούν και να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες μας. Σε κάθε τράπεζα είναι αυτό πραγματικότητα σήμερα. Αγοράζουμε λοιπόν ε, με τέτοιου είδους, με, ε, επιτόκια τα οποία ε, καθορίζουμε, συναλλασσόμαστε ώστε να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες μας μέσω αγοράς για παράδειγμα παραγόγων. Θα υφίστανται τέτοιες δραστηριότητες σε όλες τις τράπεζες. Αλλά αυτό το γεγονός δεν είναι άλοθη δεν είναι πρόσχημα για οποιασδήποτε δραστηριότητες σε όλες τις αγορές. Η δική μας ε, ε, φιλοσοφία είναι ότι όταν ένας ε, πελάτης φοβάται τους κινδύνους των αγορών και καταθέτει τις δικές του, την δική του αποταμίευση στις τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζεται σε αυτή την πράξη του. Δεν είναι το θέμα μόνο των ε, ε, καταθέσεων, αλλά η δυνατότητα δραστηριοποίησης στη συνέχεια. Τα κεφάλαια αυτά είναι ένα, ε, μια δυνατότητα απόσβεσης ή κάλυψης κινδύνων. Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί στο τι θα επιλέξουμε να κάνουμε σε σχέση με τις εμπορικές μας δραστηριότητες. Και αν υπάρχει υπερβολικός, υπερβολική εμβέλεια και δεν υπάρχει δυνατότητα να επενδύσουμε ως τράπεζες, καλύτερο είναι το πλεόνασμα αυτόν αυτό να μπορέσει να επιμεριστεί στους ε, ομολογιούχους ή μεριδιούχους, εκείνοι να αποφασίσουν πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Και τώρα με βάση την αρχή ότι ευφυείς ε, άνθρωποι θα μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδη, Μπορεί όμως ε, να είναι επικίνδυνο τέτοιου είδους δραστηριότητες να χρηματοδοτούνται με τις καταθέσεις πελατών των τραπεζών και όταν η ε, δυνατότητα παρέχεται από τους ε, συναλλασσόμενους ε, μπορεί να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη των αγορών. Το είδαμε κατά το παρελθόν ότι τεράστια τα μεγάλα κέρδη ε, μπορούν να ε, επιδοτήσουν τις εμπορικές ε, δραστηριοτήτων, τις εμπορικές δραστηριότητες τραπεζών, αλλά μπορεί και να δημιουργήσουν και κινδύνους. Προσπαθώ να είμαι ακέραιος τραπεζίτης, διότι υπάρχει μεγάλο κέρδος για την κοινωνία από αυτές τις δραστηριότητες. Αυτή η δραστηριότητα συνεπάγεται συναλλαγές στις οικονομικές αγορές και την, της, τη διαχείριση κεφαλαίων και αποθεματικών καθώς επίσης και τον καθορισμό ε, συναλλαγών ε, σε ανοιχτές θέσεις ε, ώστε να διασφαλιστεί και η ρευστότητα. Μία μεταρρύθμιση τραπεζική πρέπει να διαχωρίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Μια τέτοια μεταρρύθμιση όχι μόνο θα ενισχύσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά θα δημιουργήσει και ένα ισότιμο, ισοδίκαιο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βάρτας. Τα μέλη τώρα έχουν ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις Κάθε εισηγητή και κάθε σκιώδη εισηγητή θα έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του, λόγω του ότι πιέζει ο χρόνο, για να διατυπώσουν ερωτήσει και να πούν σε ποιον ομιλητή στοχεύει η ερώτηση. Ο ερωτώμενο θα έχει δύο λεπτά να απαντήσει. Δέκα επιπλέον λεπτά μα δίνουν οι διερμηνεί. Ελπίζω ότι θα κατανοήσετε ότι για τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές ένα λεπτό μόνο προβλέπεται, Λόγω του σχολείου του κυρίου Λάγεν θα ήθελα να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ένα μέρος του χρόνου για να εκμεταλλευτούμε με το κασλιάι με τα υπόλοιπα μέλη. Ξεκινάμε με τον εισηγητή Γκούναρ Χέκμαρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Σας ευχαριστώ πολύ. θα ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι είναι μια γενική ε, θα έλεγα συμφωνία ότι η μεγαλύτερη κίνδυνη από πλευράς εξειδικευμένων ε, τραπεζών και αυτό από την έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, φιλοξενούμενο από το δεύτερο πάνελ, συμφωνεί με αυτό ότι η μεγαλύτερη κίνδυνη είδαμε ότι ήταν σε σχέση με τις συναλλαγές λιανικής έναντι των ενυπόθηκων και στα, στεγαστικών δανείων και ποια είναι η άποψή του για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με τις ε, συναλλαγές ε, λιανικής. Υπάρχει ευρύτερη συνένεση φυσικά για ε, τη χρήση αποθεματικών. Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ απευθύνεστε, στο δεύτερο πάνελ. Μάλιστα. Ε, τότε λοιπόν ζητώ να δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση. Καθένας από εσά. Από τα αριστερά προς τα δεξιά ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Ναι, συμφωνώ πρέπει να πω ότι η δανειοδότηση για τον τομέα ακινήτων και για την ε, απόκτηση στέγης και για, την, ε, για τις οικοδομικές δραστηριότητες ε, βλέπουμε ότι αυτό υπήρξε και έναυσμα και ε, της κρίσης, όχι μόνο αυτής αλλά και προηγούμενων. Ωστόσο όμως, ε, τούτου λευθέντος δεν συμφωνώ υποχρεωτικά με το γεγονός ότι αυτό στοιχειοθετεί το ότι το πρόβλημα βρίσκεται αποκλειστικά στις τράπεζες που χρηματοδοτούσαν τέτοιες ε, δραστηριότητες δανειοδότησης, απόκτησης στέγης ή ακινήτων διότι κατά την κρίση για την ε, μετάδοση κινδύνου ήταν ο κίνδυνος ε, μέσω αυτής της δανειοδότησης και η ε, επίπτωση ντόμινο μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και με την αγορά και συναλλαγή σε παράγωγα. Δηλαδή όσον αφορά τη δανειοδότηση για την απόκτηση ακινήτων και την, τις δραστηριότητες στις security markets στενά διασυνδέονται, διότι η ε, διαμεσολάβηση αυτή ε, μεγέθυνε τους κινδύνους που απέρεαν από την ε, δανειοδότηση για την αγορά κινήτων. Όσον αφορά την άλλη παρατήρησή σας, ήδη είχα σχολιάσει προηγούμενα ότι κάθε φορά που κάνουμε λόγο για κίνδυνο για τις επιπτώσεις του διαχωρισμού δραστηριοτήτων δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι οι τράπεζες δεν είναι η μόνη ενδυνάμει ε, πάροχη των παραγόγων. Έχουμε ε, hedge banks, ε, έχουμε κάθε είδους διαμεσολαβητές που δρούν και διαμεσολαβητές που δεν είναι, διαχειρίζονται ε, καταθέσεις και όμως παρόλα αυτά παρέχουν μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό ρευστό στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι Ίσως μπορεί να μην ήταν σε καλύτερη θέση οι μεγάλες τράπεζες για να παράσχουν ρευστότητα, όμως οι άλλοι διαμεσολαβητές μπορούν να το πράξουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πήρατε τον χρόνο και των υπολείπων. Ζητώ από τους άλλους συναδέλφους το εξής. Θέλετε όλοι να απαντούν στις ερωτήσεις σας. Ένα σύντομο σχόλιο για τις εξειδικευμένες τράπεζες. Θα έλεγα υπήρξαν πρόβλημα στις ε, τράπεζες λιανικής ε, ε, και στις τράπεζες δανειοδότησης στεγαστικών δανείων. Θα έπρεπε να δούμε την δυνατότητα εξασφάλισης αυτών των συναλλαγών. Ο κύριος Γκούταρτ είπε ότι έζησε και επιβίωσε τριών τέτοιων κρίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κρίσεις αυτές στο παρελθόν μπορεί να ήταν περιορισμένου χαρακτήρα. Η μεγάλη όμως κρίση που είδαμε τελευταία είχε τέτοια εμβέλεια που είχε συστημικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να απαντήσω στι τρει αυτέ ερωτήσει. Για τι εξειδικευμένε δραστηριότητε ε, τραπεζικά, ε, όλοι συμφωνούμε ότι η πολυσχηδή δραστηριότητα, η πολυμορφοποίηση έχει ε, ρόλο κλειδιού. Για την διαχείριση ρευστότητα, ιδιαίτερα στον τομέα τη αγορά, έχει χέρια σημασία αυτό το στοιχείο. Ένα από του λόγου για το, γιατί κυβερνητικά ομόλογα αποκλείστηκαν είναι για το ότι η ρευστότητα είναι κέριου χαρακτήρα για την ε, χρήση των ομολόγων, κυβερνητικών ομολόγων. Η ισχυρή διακυβέρνηση είναι καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν ε, τέτοιες ε, κρίσεις και τέτοιοι κίνδυνοι από την νομική διαφοροποίηση δραστηριοτήτων τραπεζών. Θα ήθελα να υιοθετήσω την άποψη ότι η χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων υπό το ακαδημαϊκό πρίσμα αληθεύει ότι η ασυμμετρία ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξειδικευμένες τράπεζες που έχουν πολύ στενή σχέση με τους πελάτες τους αυτούς είναι οι καλύτερες και πιο ενδεδειγμένες να μειώσουν αυτή την ασυμμετρία στην πληροφόρηση και ενημέρωση και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ώστε να είναι πιο ε, κερδοφόρες ε, και πιο εγγυημένες οι δραστηριότητες ε, που ακολουθούν έναντι των πελατών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρώτος σκιώδης εισηγητής Γιάκοπ Φον Βάιτσεγκερ. Θα παρακαλούσα να περιοριστείτε σε ένα λεπτό και ερωτή, ερώτηση να διατυπώσετε που μπορεί να απαντηθεί σε δύο λεπτά γιατί έχουμε 20 λεπτά όλα όλα για όλους τους σκιώδεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για τον καθηγητή Μάρκο Παγκάνο όσον αφορά την έκθεση στην οποία αναφέρθηκε για το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Στην έκθεση αυτή αποδεικνύεται αυτό το οποίο προσμετράται ως κοινωνικό κόστος ε, των τραπεζών, αυξάνεται με το μέγεθος της τράπεζες και ε, μέσω και της αυστηρότητας προσβεί δανειοδοτικές δραστηριότητες. Ε, χρησιμοποιείται ως παράμετρο το, τη δανειοδότηση σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού. Και η ερώτησή μου προς εσάς είναι κατά πόσον θεωρείτε ότι αυτή η ε, παράμετρος δάνειο ε, διανοδότηση προς τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην μεταρρύθμιση των τετραπεζών για να αξιολογήσουμε κατά πόσον θα πρέπει να γίνει διαχωρισμό σε κάτι ή όχι. Ναι, μια σύντομη απάντηση να σας δώσω ναι, όντω θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη παράμετρο αυτή, κατά πάσα πιθανότητα σε συνδυασμό με άλλε. Ε, διότι, προκειμένου να απαντήσω πλήρω στην ερώτησή σα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε άλλε αντίστοιχε παραμέτρου, όπω για παράδειγμα το ε, ε, κατά πόσον υπάρχει συμμετοχή σε εμπορική δραστηριότητα, διότι η μη διανοητική δραστηριότητα δεν είναι μόνο εμπορικέ δραστηριότητε, αλλά μπορεί να είναι και άλλε δραστηριότητε, οι οποίε θα μπορούσαν και αυτέ να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ναι, ε, με κάποιε διαβαθμίσει βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Καμάλ από το ECR, αλλά έχει αποχωρήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι κάποιο άλλο εδώ που να τον αντικαθιστά. κανεί, επομένω, περνάμε ευθεία στου ουλελευθέρου. Η Σίλβη Γκουλάχ, παρακαλώ. Μία σύντομη ερώτηση και πάλι. Ποια είναι το στρατηγικό σα όραμα, ρώτησα και προηγουμένω, πώ θα χρηματοδοτήσουμε την Ευρωζώνη και την Ευρώπη με ανεξάρτητο τρόπο στα επόμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι μέσω διαστροτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να γίνει, μέσω καλύτερης εποπτείας, μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου ε, ο ρόλος και του μηχανισμού εξυγίανσης θα μπορούσε να βοηθήσει. Ε, σε ποιον απευθύνεται το ερώτημά σας? Προς το Finance Watch, δεδομένου ότι έχουμε την τιμή να έχουμε και μία γυναίκα εδώ σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον πάνελ. Ευχαριστώ πολύ θα έλεγα ότι εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, χρειαζόμαστε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος. Και όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, θεωρώ ότι οι συστημικοί κίνδυνοι απορρέουν από πολύ μεγάλη εμπορία, κυρίως εμπορία παραγόγων και κάτι το οποίο, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καταστροφικό για την πραγματική οικονομία ε, τι θέλουμε να προλάβουμε. Θέλουμε να μην έχω μια άλλη κρίση σαν αυτή που βιώσαμε προηγουμένως. Και θα ήθελα να επανέλθω απευθείας ε, σε αυτό που είπε ο κύριος Γκούτχαρτ. Αν δούμε τη σχέση μεταξύ ΑΕΠ και της ε, ανάπτυξης του ΑΕΠ. Στην τελευταία κρίση το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε έξι φορές το ΑΕΠ του ε, και δεν θα αναφέρω καν τα ποσοστά ανεργία σε άλλες χώρες. Ο συστημικός κίνδυνος λοιπόν και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα θα πρέπει να είναι οι στόχοι μας προκειμένου να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φιάμπιοντε μαζί από, τους, ε, από την ΚΟΕ. Ερώτηση για τον κύριο Παγκάνο. Αναφέρθηκε στην έκθεση ε, η σχέση ε, δανείων ε, χρέους και η δυνατότητα αγοράς από υπηρεσιών από εξειδικευμένες τράπεζες αν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότηση από την αγορά. Έτσι το χρηματοδοτικό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξηθεί πολύ και πόσο ε, πιθανή είναι η χρηματοδότηση από την κεφαλαία αγορά αυτών των επιχειρήσεων. Αυτή ήταν για τον κύριο Παγκάνο. Ο κύριος Παγκάνο θα απαντήσει. Θέλω να πω ότι η χρηματοδοτική ροή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμποδίζεται πολύ σήμερα από ένα μεγάλο παίκτη στις χρηματοοικονομικές αγορές, κυρίως στις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Ένας βασικός τρόπος επανενεργοποίησης της ε, δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ειδικότερα που μας ενδιαφέρουν πολύ είναι οι κυβερνήσεις να ε, μειώσουν αυτό το crowding out που γίνεται πολύ τώρα στις ε, χρήματα αγορές και κάποιες ε, χώρες της περιφέρειας. Ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λάμπερτ, Χιώδης των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση και σχόλιο προς τον κύριο Κρέμα από την Μπεβεβέρ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, είχαμε τον ίδιο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Είναι σοφή η συμβουλή σας στο Κοινοβούλιο να σταματήσουμε αυτή την πρωτοβουλία και να σώσουμε ενέργεια για να την έχουμε για καλύτερο σκοπό. Αυτό το κάνετε για να σωθεί η οικονομία. Είναι ευπρόσδεκτη η συμβουλή του τραπεζικού τομέα. Έπρεπε να σας έχουμε, έπρεπε να σας έχουμε ακούσει περισσότερο. Θα αποφεύγαμε τη μεγάλη καταστροφή του 2008 που μάλλον δημιουργήθηκε από την ανοησία των πολιτικών. Ο παρακαθήμενός σας είπε και έδειξε ότι μπορείτε να προσφέρετε κάθε είδους υπηρεσία στους πελάτες και στο τέλος να διατηρήσετε ε, κανένα κίνδυνο και ανοιχτές θέσεις στον ισολογισμό σας. Γιατί έχετε κάνει ε, ε, προστασία από επενδυτικές τράπεζες. Αυτό αν γίνεται για την Βαν Μπρέντα, γιατί να μην γίνει για σας. Και αν τώρα μπορείτε να δώσετε υπηρεσίες με επιδοτούμενο κόστος, εγώ είμαι φιλελεύθερος της αγοράς και θα ήθελα οι πελάτες να πληρώνουν το πραγματικό κόστος, όχι να επιδοτείτε το κόστος λόγω των φορολογουμένων. Με ενδιαφέρον θα ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Πρέπει να πω ότι δεν έχω ε, τη σωστή απάντηση. Κάποια στοιχεία θα πω σχετικά με το πώς οι γενικές τράπεζες μπορούν να προσφέρουν λύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δομή hedging των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι περίπλοκη γιατί οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι σύνθετοι. Δεν είναι μόνο θέματα ανιοδότησης των ΜΜΕ, είναι πολλές υπηρεσίες μεγάλης εμβέλειας που είναι θεμελιώδης για τις ΜΜΕ για να αποφύγουν την μεταβλητότητα των κερδών ή κινδύνους που δεν θέλουν να αναλάβουν. Οι, όλες οι συναλλαγές, όπως είπε ο κ. Βάουτερ, δεν είναι τόσο εύκολες ε, ε, όπως ας πούμε η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Κάποια ιδρύματα ε, κάνουν εξαγωγές στο Μεξικό και θα πρέπει να καλυφθούν από άλλα μέσα γιατί τα clearing house στην Ευρώπη δεν καλύπτουν τον κίνδυνο από το μεξικανικό πέσος. Ε, οπότε πώς θα δώσουν αυτές τις υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές. Η λύση που βλέπει η πρόταση είναι να ε, υπάρχουν δύο διαφορετικές μονάδες τραπεζικές που δίνουν δύο διαφορετικά προϊόντα. Τεχνικά γίνεται αυτό. Αλλά από άποψη κόστους ωφέλους δεν έχει νόημα. Δεν, ε, εν μέρη απάντησα στη σύνθετη ερώτηση, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Ε, σχέση κόστος ωφέλους για τον ε, φορολογούμενο. Ε, υπέρ της οικονομίας δρούμε. Σε τελευταία ανάλυση θέλουμε να προωθήσουμε την οικονομία. Ο τελευταίος σκιώδης απόψε, ο Μάρκος Σάντι από τη FTD. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον καθηγητή Παγκάρνο το εξή, διότι δεν μου απαντήθηκε πριν για τα παράγωγα. Αν εντό μια ε, ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματο θεωρείται ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα μέσο αξιολόγηση, ένα ανεξάρτητο μέτρο ε, αξιολόγηση του κινδύνου των παραγόγων για τι πιο μεγάλε τράπεζε, όπω έγινε στι ΗΠΑ το 2008. Και μια δεύτερη ερώτηση ε, και πάλι για το πώς βλέπετε το ρόλο στο μέλλον για το crowdfunding ως νέο τρόπο ε, χρηματοδότησης και νέο ε, μέσο διαφοροποίησης του κινδύνου ε, για τις τράπεζες, του πιστοτικού κινδύνου των τραπεζών. Δηλαδή να μετατοπιστεί ο κίνδυνος για τις τράπεζες σε αυτό το μέσο, εάν στο μέλλον βέβαια φτάσει και σε ε, σημαντικές διαστάσεις. Για να εξοικονομήσουμε και χρόνο να σταθώ στην πρώτη ερώτηση, στα παράγωγα. Όντως, ε, τα μεγαλύτερα και τα πιο επικίνδυνα ε, στοιχεία ε, για τις τράπεζες είναι όντως από τις αγορές παραγόγων. είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τους κινδύνους αυτός, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο οι πολύ μεγάλες τράπεζες μπορούν να ε, τηρούν τέτοιες στάσεις και έχουν και κίνητρα προκειμένου να δρουν κατά αυτόν τον τρόπο είναι διότι ε, τα ιδρύματα με τα οποία εμπορεύονται θεωρούν ότι είναι ασφαλέστερα από άλλους πιθανούς εκδότες ε, παραγόγων διότι ακριβώς απολαμβάνουν αυτή την εγγύηση του too big to fail, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν. Και ίσως ε, το πρόβλημα αυτό ε, θα μπορούσε να είναι ε, μικρότερο και δεν είναι να μην είναι τόσο παρεμβατικό, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον αυτή η εγγύηση του big to fail από τράπεζες οι οποίες πραγματικά στοιχηματίζουν στις αγορές παραγόγων μέσω αυτής της εγγύησης του too big to fail που τους βοηθά θα μπορούσα να προσθέσω και το εξή. Υπάρχει και το πλαίσιο το οποίο υποχρεώνει τις τράπεζες να περνάνε από το CCP, κυρίως ε, μεγαλύτερες τράπεζες, ή ε, τι, τεχνικές μετριασμού του κινδύνου, ε, που είναι αυτό το οποίο ε, κυρίως κάνει το τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι λόγω πειθαρχία, τώρα πλέον υπάρχει χρόνος για μία επιπλέον ερώτηση ΚΑΤΣΔΙ πριν δώσω το λόγο ε, στον Κούναρ Χέκμαρ. Ξέρετε ότι ο συνάδελφος Κέλλερ ζήτησε να υπάρχει διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος. Είναι η Ναγκίλ. Η συγγήτρια για τα αμοιβαία κεφάλαια Θα ήθελα να λάβω το λόγο στο πρώτο τμήμα στην πραγματικότητα, γιατί ο καθηγητής Χέλουικ, ε, ε, δεν ξέρω αν είναι εδώ, είμαι η συγγήτρια για τα αμοιβαία ε, κεφάλαια και θα ήθελα ε, να ακούσω, δεδομένου ότι ήσασταν, πολύ επικριτικός και σε κάποιες περιπτώσεις δικαίως και εμείς προσπαθούμε να αναζητήσουμε έναν τρόπο να διασκεδάσουμε αυτή την, την ανησυχία, το, ε, την άποψή σας. Η SEC έκανε πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση τον Ιούλιο και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη ΣΥΠΑ. Επίσης θα ήθελα... Ε, επειδή ανησύχησα πολύ, ε, διότι την περασμένη εβδομάδα στις Financial Times, στην πρώτη σελίδα, διάβασα ότι ε, κάποιες από τις μεγαλύτερες σταθερές ΚΑΕ λόγω των μεταρρυθμίσεων στα αμοιβαία κεφάλαια ε, σκέφτονται να συστήσουν ε, ιδιωτικά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία θα είναι εκτός ε, δικαιοδοσίας και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ουσιαστικά αυτό έρχεται να προσθεθεί στα αυτό που έλεγε ο καθηγητής Γκούτχαρτ, ότι το πρόβλημα και ίσως και καλό στοιχείο του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ότι είναι πολύ καινοτόμοι, αλλά μάλλον είναι καινοτόμοι ε, με λαθασμένο τρόπο, προσπαθούν να βρουν τρόπο ε, ώστε να μην ε, τους ελέγχει κανείς. Ε, πώς βλέπετε αυτή την προσέγγιση για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και κυρίως για τον ευρωπαϊκό τομέα στο σύνολό του. Ευχαριστώ Νίνα. Νομίζω ότι η αίσθηση κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μην αυταπατώμεθα. Ε, πολλά τα μία και κεφάλαια ε, ε, ενέχουν τον κίνδυνο ε, της απόσυρσης των καταθέσεων. Ε, και αυτό είναι ε, κάτι αυτό είναι ένα, ε, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει συντονισμός από τους επενδυτές. Τώρα, ένα ανοιχτό φαντ το οποίο επενδύει σε στοιχεία που δεν είναι ε, αμεσαρευστά, ε, πάλι ενέχει τον κίνδυνο του ραν. Εμείς έχουμε και άλλα ταμεία εκτός από τα, τα χρηματοοικονομικά. Πάντα ενέχουν συστημικό κίνδυνο. Τώρα, το πρόβλημα που έχω με το αμερικανικό σύστημα είναι ότι το SEC που είναι υπεύθυνο, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, θεωρεί ε, σκέφτεται πάντα την προστασία των επενδυτών και όχι του συστήματος. Και υπ' αυτή την έννοια δρά πολύ διαφορετικά, έχει διαφορετική αντίληψη από τους τραπεζικούς επόπτες και γι' αυτό μεταξύ άλλων κολλησιεργούν ως προς το θέμα αυτό τόσο πολύ καιρό. Ευχαριστώ κύριε Χέλβικ. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή Γκούναρ Χόκμαρ για να κλείσει, θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που μας έδωσαν 10 ακόμη λεπτά. Ευχαριστώ και εσάς που με τη πειθαρχία σας ε, μας επιτρέψατε να τηρήσουμε το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, ιδιαίτερα τους αποψινούς μας προσκεκλημένους που συνέβαλαν με τόσο διαφοροποιημένο και ενδιαφέροντο τρόπο. Γκούναρ για το κλείσιμο. Ευχαριστώ και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου γιατί ήταν πολύ καλές οι παρουσιάσεις, πολύ καλά προετοιμασμένες ε, για μας ε, και πολύ θετικές. Δεν θα προσπαθήσω να παρουσιάσω πολλά συμπεράσματα γιατί ο κίνδυνος ε, είναι να διαφοροποιηθούμε στις απόψεις μας και δεν θέλω, γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και θέλω πνεύμα ενότητας. Ε, υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά τα οποία θα συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί τώρα πήραμε τροφή για σκέψη. Καταρχήν, τι γίνεται ως καταθέτες εξαρτώμεθα περισσότερο από εξειδικευμένες τράπεζες και τι γίνεται με τη διαδικασία Βερολίνου. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με την δημιουργία ρευστότητα όταν έχουμε περισσότερες ειδικέ τράπεζες. Πολλοί συνάδελφοι κάνουν ανοιχτές συγκρίσεις με τις ΙΠΑ, αλλά η τραπεζική δομή στις ΙΠΑ αποτελεί αποτέλεσμα εξελίξεων 100 ετών, όπως στην Ευρώπη. Τι γίνεται με τη δημιουργία ρευστότητα και τι γίνεται με τους συστημικούς κινδύνους όταν εξαρτώμεθα περισσότερο από εξειδικευμένες τράπεζες. Αν δούμε στο παρελθόν και θυμηθούμε και παλιές συζητήσεις, ε, θα δούμε ότι υπάρχουν ερωτηματικά που κάποιοι τα είδαν επιφυλακτικά όταν τα έθεσα, αλλά νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμά μου είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Γιατί θα πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο σταθερό πλαίσιο γίνεται. Αλλά και αυτό είναι ένα παράδοξο. Όσο γίνεται πιο δυναμικό επίσης. Δηλαδή σταθερό πλαίσιο και δυναμικούς ε, παράγοντες της αγοράς. Αυτό πρέπει να συνδυάσουμε. Ευχαριστώ πάλι τους προσκεκλημένους μας τους συναδέλφους, τον πρόεδρο και τον προηγούμενο ε, πρόεδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.